Bene, colleghi, abbiamo molto lavoro da fare. Cominciamo su. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά στην ημερησία διάταξη. Ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Ah, Θέλω να βάλω απλώς ένα θέμα... Yes, please. Θέλω απλώς να βάλω ένα θέμα διαδικασίας. Καλημέρα σας. Οι λίστες ψηφοφορίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήρθαν ψες αργά το βράδυ, ίσως και μετά τις 10. Οι άνθρωποι που έπρεπε να δουλέψουν ήταν ήδη πάρα πολύ αργά και πολλοί από αυτούς φυσιολογικά εκτός γραφείων. Θεωρούμε ότι ήταν σωστό να αναβληθεί η ψηφοφορία για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, και άλλοι έκαναν αυτή την παρατήρηση. Ο Χάουιτ. Η, η πλειοψηφία θα αποφασίσει. Κοιτάξτε, είναι γενικότερο το θέμα. Να πω για τα πρακτικά. Πρώτον, Υπάρχει μία μόνο συμβιβασμό. Αν θυμάστε τη συζήτηση που έγινε χθε το πρωί, ε, είχαμε πάνω κάτω καταλήξει και όλα είχαν τελειώσει χθε τη μία το μεσημέρι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το προσωπικό δεν μπόρεσε να φέρει πέρα σε μπάση περιπτώσει τι διαδικασίε από εκεί και πέρα. Έπρεπε η γραμματεία να μας βοηθήσει να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε σήμερα το πρωί. Αν υπάρξει αναβολή για την επόμενη εβδομάδα, θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να είναι η πρώτη ε, ψηφοφορία που θα γίνει, γιατί το απόγευμα θα πρέπει να φύγω. Νομίζω ότι εμείς σαν μέλη κάναμε ό,τι μπορούσαμε και το κάναμε σε σωστό χρόνο. Και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ήταν ιδιαίτερα ευέλικτοι χρονικά και δεν είχαμε πολύ χρόνο αλλά τα καταφέραμε και θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα γιατί τίθενται τέτοιου είδους θέματα. Αλλά αν αναβληθεί θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, γιατί θα πρέπει την τρίτη απόγευμα εγώ να φύγω. Σαλαφράγκα. Gracias, señor presidente. Eh, yo lo que quiero decir es que me parece poco serio y poco profesional. Φαίνεται ότι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι πάρα πολύ επαγγελματικό, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση και μιας και έχουμε ολοκληρώσει εμείς την προσπάθεια που έπρεπε να ολοκληρώσουμε σαν βουλευτές, να μην προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Εγώ πήρα ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια της νύχτας ε, λέγοντας ότι θα γίνει ψηφοφορία την επόμενη Τρίτη. Ενώ τώρα το πρωί εδώ έρχομαι και μαθαίνω ότι η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το πρωί. Δεν καταλαβαίνω. Ε, δεν μπορούμε να αναβάλουμε, να ξαναβάλουμε. Τέτοιου είδου σε πάση περιπτώσει, αστάθεια δεν είναι δικαιολογημένη. Εφόσον υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ψηφοφορία σωστά, αν κάποιες πολιτικές ομάδες, σε πάση περιπτώσει, το πιστεύουν αυτό, εγώ δεν είμαι κατά της αναβολής για την επόμενη εβδομάδα πάντα. Αλλά προσωπικά εγώ προτιμώ να ψηφίσουμε σήμερα. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Τάνοκ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε σαν ομάδα των συντηρητικών. τελευταία στιγμή δεν είναι σωστό να δημιουργούνται τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνη σε οποιονδήποτε, αλλά νομίζω ότι μια και ο εισηγητή θέλει να περάσουμε σε ψηφοφορία, νομίζω ότι υπάρχει συνένεση. Υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον για να γίνει ψηφοφορία σήμερα το πρωί νόμο των Φιλελευθέρων, συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε πως υπήρχαν πρακτικά προβλήματα και βεβαίως καλό θα ήταν να μην ε, είναι έτσι η κατάσταση, αλλά νομίζω πως το καλύτερο είναι να τιμήσουμε τον εισηγητή και τους ανθρώπους που εργάστηκαν με μεγάλη ευελιξία μέχρι την τελευταία στιγμή. Ε, γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ του να ψηφίσουμε. Πέρα λοιπόν από την καλή θέληση όλων, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο περιορίζει αν θέλετε την διαθεσιμότητα του τελικού κειμένου και εμποδίζει λίγο τη δυνατότητα λήψης απόφασης. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι τι γίνεται με την πλειοψηφία. Οι φιλελεύθεροι, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι συντηρητικοί και οι σοσιαλιστές οι αρχηγοί του ενώ, ε, ζήτησαν να υπάρξει ψηφοφορία σήμερα. Οπότε εγώ απλά θα υπακούσω στην θέληση της πλειοψηφίας και θα προχωρήσω στις ψηφοφορίες. Επαναλαμβάνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξανασυμβεί στο μέλλον. Καλώς λοιπόν θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες για το Αζερβαϊτζάν και για τη συμφωνία. Παράγραφος 1, τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Δεκτή. Ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα λέω όλα κάθε φορά, λέει ο πρόεδρος. Περνάω τώρα στην τροπολογία 39. Α, όχι, έχει καταπέσει. Η συμβιβαστική 2, τη συμβιβαστική 2 θα ψηφίσουμε τώρα σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα της δύο ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα της δύο ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Περνάμε στη συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 44. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται. Αν θέλετε έλεγχος ηλεκτρονικά για τη 44. Έλεγχος ηλεκτρονικά για την 44 επαναλαμβάνει ο, ο πρόεδρος. 44. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 50. Ποιοι είναι υπέρ της 50 παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απορρίπτεται. 51. ή μάλλον όχι, διορθώνει ο πρόεδρο, διακόπτει μια στιγμή. Επιστρέφουμε στο 50 γιατί έχει ζητήσει ηλεκτρονικός έλεγχο ε, της 50. Ε, ε, Επανερχόμαστε παρακαλώ ψηφίστε για την 50. Την 50 λέει συνέχεια ο πρόεδρος. Oh. 007. Όσοι δεν ψηφίσατε παρακαλώ να ψηφίσετε τώρα πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται η 50. Περνάμε στην 52. 52. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54. Ποιοι είναι υπέρ. Α, συγγνώμη. 53. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 54 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. 58 και 59 από κοινού, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 60 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές Πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. 61 τώρα. Κόβατσεφ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 62 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά. Είναι απαραίτητο να υπάρξει έλεγχο στην 63. Manca un voto. Chiudiamo la votazione. Κλείνω την ψηφοφορία. Ε, για την 64 θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 65 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 66 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 4 τώρα, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. 71, όχι, συγγνώμη, 72 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Από την 73 μόνο το δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε τώρα στο 76 και εδώ ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα, συνάδελφοι, ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο 89. Το πρώτο τμήμα του 89 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Το πρώτο τμήμα του 89. Το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά Ποιοι απέχουν απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 92, το οι προηγούμενες έχουν καταπέσει. Λοιπόν. Α, κάποιος θέλει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της 89. Ζητήθηκε λοιπόν ο ηλεκτρονικός αυτός έλεγχος. Ψηφίζετε παρακαλώ. δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία. Όπως λέει ο συνάδελφος Πάσκου. 92 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο 93. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια ψηλά γιατί δεν καταλαβαίνω λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος τώρα της 94 δεκτή η 94. Περνάμε τώρα στην 99. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φαινότανε, δεν χρειάστηκα έλεγχος, αν και κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν σαμποτάζ. Φτάσαμε στην 100, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η 100. 101. 102, συγγνώμη. Και είναι υπέρ της 102. Κατά. Αποχές. Δεκτή η 102. 104. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 105. Ψηφίζουμε. πέραση ψηφοφορίας δεκτή. Περνάμε στο 107. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται η 107. 108. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτό. 109. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 τώρα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 113 Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 114. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στην 120 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 τώρα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 128 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 128 δεν είναι ξεκάθαρο. Τρεις συνάδελφοι πρέπει να ψηφίσουν. Δεκτή. 129 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 130 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 131 αποσύρθηκε, η 132. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα περνάμε στην 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, απορρίπτεται. 13, συμβιβαστική 13, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η 13. 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 17, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 18, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 19, πολύ σημαντική 19 λέει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, όχι, απέχουν δεκτή. Ακόμα και αυτή έγινε δεκτή. 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Για την 24, Watson. Υπάρχουν τρεις συνάδελφοι που δεν ψήφισαν ακόμα. Ψήφισαν κλείνει η ψηφοφορία δεκτή η τροπολογία. Περνάμε τώρα στην 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τι θέλετε. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος επιμένετε. Μάλιστα, θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 25. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Η δημοκρατία σημαίνει το να υπακούει κανείς τις επιθυμίες των άλλων. Λοιπόν, 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στο 35 βίγγενιν υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 1 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3 και 4 τα Τάνο πιανάκου ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 8 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 9 υπέρ, κατά, και απέχον δεκτή. Η 10 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή και η 10. Τώρα πλέον θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου όπως τροπολογήθηκε. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα, ένας δεν έχει ψηφίσει, τέλος της ψηφοφορίας, δεκτή. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ωραία, περνάμε στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία για να είμαστε πιο σύντομοι και αρχίζουμε αμέσως τις ψηφοφορίες.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 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 και 46, 46 και 47 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54-55 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 56. Ε, όχι. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστή. Διακόπτε ο πρόεδρος. Λοιπόν, μιλάμε για την τροπολογία 66. Ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 68, δεύτερο τμήμα μόνο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Facciamo un check. έλεγχος. Αν κερδίσω εγώ, Κερνάω σαμπάνια σε όλους. Τριάντα ένα υπέρ. Εξήντα εννέα τώρα, υπέρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν τα ίδια ε, με την προηγούμενη έκθεση. Νομίζω ότι ψηφίσαμε με έναν τρόπο στη μια έκθεση και αντίστροφα στην άλλη για το ίδιο θέμα. Αν θυμάμαι καλά. Πάντως νομίζω πως εκεί δεν κάναμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ε, ε, Κοιτάξτε, το ίδιο είπαμε. Εγκρίνονται και τα δύο. Δεν υπήρξε διαφορά. Εγκρίθηκαν και τα δύο. Έχουμε το έγγραφο μπροστά στα μάτια μας. Αφού δεν με πιστεύετε να σας το επιβεβαιάσει και η γραμματεία. Στην 76 για το Αζερβαϊτζάν το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε και έχει ακριβώ την ίδια διατύπωση 68, με την 68 αυτής εδώ της έκθεσης το δεύτερο τμήμα που είναι Ακριβώς η ίδια διατύπωση. No, eh, eh, dal momento che il notaio ha detto così... Κοιτάξτε, αφού εδώ συμβολογράφος μας ε, είπε πως εγκρίθηκε, ε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, είμαστε στην τροπολογία 69 τώρα, συμπιστρέψουμε στην ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73. Όχι, 74 γιατί καταπίπτει η 73. 74 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε- allora, chiedo, chiedo, allora, si può chiedere la verifica del numero legale, però i... Εγώ να ζητήσω επαλήθευση ηλεκτρονική. Αλλά οι απόψει σα που φτάνουν από εδώ και από εκεί δεν ε, μπορούν να ληφθούν υπόψη. Μπορείτε να ζητήσετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Το μόνο. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό που έχω για το διοικητικό σκέλος, ε, για τους διοικητικούς υπαλλήλους μας, βρίσκω πως δεν έχουν καμία δουλειά να δίνουν τη γνώμη τους για τις ψηφοφορίες που έγιναν ή που γίνονται ή για τις τροπολογίες. Και εγώ το ίδιο υπογράμμισα. Εσείς ζητήσατε επισήμως ηλεκτρονικό έλεγχο για την 78. Μάλιστα. Ωραία. 78. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 80. Τροπολογία 80. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Γιατί πολύ λίγα χέρια σηκώθηκαν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την, για την ε, τροπολογία 80. Τρεις συνάδελφοι δεν ψήφισαν ακόμα. Ψήφισαν τέλος ψηφοφορίας. Ε, τα βλέπετε εδώ. Σαμποτάζ μου κάνετε. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Κοιτάξτε, σα παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σα. Γιατί αν σηκώνετε ένα-δύο χέρια από τη μια και ένα-δύο χέρια από την άλλη, ε, δεν μπορούμε να προχωρά, ε, προχωρήσουμε. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 82. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ο 90 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 90. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 92. Παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Έγκρινεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Εδώ πρέπει να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό. Vi prego di όλοι.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 108 υπέρ κατά αποχές όχι, ελάχιστη. Ελάχιστη σηκώσατε τα χέρια σας. 108 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ancora due colleghi. Chiudiamo la votazione. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. 109. Si diverte molto il collega Galler. Ωραία τα περνάει ο Γκάλερ. Άμα όμως σήκωνε και το χεράκι του θα ήταν καλύτερα. Το νόβι, και favorevole? 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 10. Υπέρ. Όχι. Η 11 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 10. Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε. 11. Υπέρ ποιοι είναι, κατά. Αποχές. Ελέγχουμε, γιατί δεν κατάλαβα. Για την 11, για την 11 ψηφίζουμε. Chiudiamo la votazione. Τέλο τη ψηφοφορία. Έκρινεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. απόχέ. Έγκρινεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Allora passiamo al 25. Favorevoli. 25 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση τώρα για το 25 ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25 Τέλο Τέλος της ψηφοφορίας. Καλά έκανα και ζήτησα έλεγχο, εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος Τροπολογία 4. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την έκθεση. Όποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ να πατήσουν το πράσινο. Mancano due colleghi, chiudiamo la votazione. Sì. Va bene, approvato. Adesso passiamo al grosso Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε, αφού εγκρίθηκε αυτή η έκθεση, στην ψηφοφορία της έκθεσης Howitt. your σας παρακαλώ να συνεργαστείτε σηκώνοντας τα χέρια σας ε, για να μπορέσουμε να το, τελειώσουμε γρήγορα. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Μήπως μπορείτε να μας σερβίρετε καφέδες. Είδα ότι γυρνάνε οι καφέδες απ' έξω και δεν έρχονται εδώ αλλά η καφέινη μας πέφτει. Πέφτει με τις ψηφοφορίες και είναι επικίνδυνο. Ε, Δέχομαι την πρότασή σας. Εγκρίνεται, αλλά λείπει ο καφές. Μας λείπει. Λείπει ο καφές. Πρέπει να περιμένουμε λίγο να φέρουν. Ο κύριος Χάουιτ θέλει το λόγο. Ε, συμφωνώ πλήρως με τον ε, κύριο Βανόρντεν, αλλά σε καθαρά διοικητικό επίπεδο νομίζω πρέπει να έχει ενημερωθεί η γραμματεία και μου ζητούν να το πω. Η παριθμόν 78 του κυρίου Κράισλερ Ντόρφλερ έχει αποσυρθεί. Η συμφωνία στη... επί της έκθεσης του Γκράχαμ Βότσον για τις κυρώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται στις ε, προφορικές τροπολογίες, αλλά ε, είχε συμφωνηθεί και θέλω να το θέσω αυτό και μου είπε η γραμματεία πως δεν έχουν βάλει τις τροπολογίες με βάση τη σειρά της ψηφοφορία. Οπότε μου είπαν να σας ζητήσω να ξεκινήσετε με τις προφορικές τροπολογίες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 εγώ απλώς διαβίβασα αυτό που μου είπε η γραμματεία. Αν τώρα λένε κάτι άλλο, εντάξει. Ναι, Ωραία, ξεκινάμε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Ναι, ναι, ναι, εγκρίθηκε, σαφώς. Αλλά αφού επιμένετε, εντάξει, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεύτερο τμήμα της 1, της συμβαστικής 1. Συνάδελφε Γκάλερ, παρακαλώ. Δεν ακούμε οι διερμηνείς. Ψηφίσαμε, ναι. Λείπουν λοιπόν, τρεις όμως. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ο κύριος, ε, ο συνάδελφος Γκάλερ είναι που μου πάει κόντρα. Λοιπόν, περνάμε στο 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38. Όχι, περνάμε στη 40 γιατί γκρίθηκε η συμβιβαστική. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42-43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές θα έκανα μια επαλήθευση εδώ Γιατί 51 51 ηλεκτρονικός έλεγχος Λείπει ένα συνάδελφο που δεν ψήφισε. τέλο ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28-28. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 χωριστή ψηφοφορία υπέρ πρώτο τμήμα συγγνώμη ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πεν, όχι, 64, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελάχιστα είναι τα χέρια που σηκώνονται και εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 66. Voto elettronico. Aperta la votazione. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. Να επαληθεύσουμε. Για την 72 η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, κάποιοι να ψηφίσετε παρακαλώ τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 όχι έχει αποσυρθεί 78 και αυτό έχει αποσυρθεί ωραία 80 υπέρ όχι μισό λεπτό μισό λεπτό 81 ψηφίζουμε τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ο συνάδελφος Πάσκου θέλει ηλεκτρονικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ναι, για την 99. Για την 99 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, δύο συνάδελφοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 105. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Είμαι πιο ήσυχο όταν έχουμε κάνει ηλεκτρονικό έλεγχο. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, Τρία χέρια όλα και όλα σηκώσατε. Ας ξαναψηφίσουμε 116 υπέρ, κατά. Ε, τώρα εγκρίνεται, ναι, σαφώς. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εντάξει, ευχαρίστω να το επαληθεύσουμε. Λείπουν κάποιοι συνάδελφοι. Ωραία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία, λέει ο κύριος Πάσκου δίπλα. Λοιπόν, 121 υπέρ. υπέρ κατά εγκρίνεται. 122 ε, σε κατά τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 131. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω αν εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αφού είναι δική μου η τροπολογία, θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 133 ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Α, υπάρχει όμως πρώτα η προφορική τροπολογία μαζί με την συμβιβαστική οκτώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Περνάμε τώρα στην 143. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται μου φαίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 143. Va bene, allora votate Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Bene, chiudiamo la 145. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ θα χρειαστεί ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 145. Ψηφίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πέρα στις ψηφοφορίες. λοιπόν, 147-148 από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 149 υπέρ. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 147-148 λοιπόν. Ψηφίστε. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Τέλος. Σαφώς γίνεται δεκτή. Η 47-48. 149 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά τις 149. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 151 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ, α, εδώ υπάρχει και προφορική τροπολογία στην 152. Λοιπόν, 152 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 153, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 153. Κυρία Κοπά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία. Η 154 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 155. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 158 υπέρ. Και είναι υπέρ της 158 κατά αποχές δεκτή. 159 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 165. 165 τώρα. Βερζιά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Ποιοι είναι υπέρ 166 ποιοι είναι υπέρ κατά Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη, 166, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Δεν θα το ξανακάνω το λάθος. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβιβαστική 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. 169. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 170 υπέρ. Κατά. αποχές δεκτή Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 14, πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό και το δεύτερο τμήμα. «182» της κυρίας Βερζιά, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. «184» υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 Θέλετε να υπάρξει λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για την 184. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Λοιπόν, μεγάλη πλειοψηφία. Συμβιβαστική 15. Με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 193. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για την 193. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. παρακαλώ να βοηθάτε σηκώνοντα ψηλά τα χέρια σας γιατί αλλιώς προσπαθώ να κρίνω από τους 4-5 που το κάνουν μόνο. Δεν θέλω να φανώ, να προδώσω την εμπιστοσύνη σας. Συμβιβαστική 17. Διορθώνει ο πρόεδρος, διορθώνει. Όχι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 194. Ποιοι είναι υπέρ τώρα. Κατά. Συμβιβαστική 17. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. 198. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. 200. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 18 με προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα. είμαστε κατά της ε, προφορικής αυτής τροπολογίας γιατί αφορά τις εκτελέσεις στην ε, Λευκορωσία και εμείς επιμένουμε σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι η Λευκορωσία η μόνη χώρα με εκτελέσεις. Δεύτερον, η τραγωδία αυτή η οποία ήταν πραγματικά σοκ για εμάς συνέβη την Παρασκευή που μας πέρασε. Δεν έχει σχέση με το 2010. Ευχαριστώ. Sí, um, I'm, Λυπούμε που το ακούω γιατί προφανώ το είχαμε συζητήσει στην συνάντησή μα και είναι σαφέ αν υπάρχει αντίρρηση δεν μπορεί να ψηφιστεί. Απλά θέλω να πω προ τον κύριο Σιμπ και του συναδέλφου του ΕΛΚ ότι εγώ προσωπικά ω συζητητή υποστηρίζω την ε, τροπολογία του και να του στηρίξω να τη φέρουν και στην Ολομέλεια. Σεβαστή η θέση των φιλελευθέρων αλλά είναι σωστό αυτό το οποίο κατέθεσε το ΕΛΚ. Και θα υποστήριξω μία τροπολογία στην Ολομέλεια για να μπει στο τελικό κείμενο. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Θα δούμε αν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει για την Ολομέλεια μια συμφωνία. Καλώς. Τώρα για τη συμβιβαστική 18 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το δεύτερο τμήμα της 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Περνάμε τώρα στην 203. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 204. Ποιοι είναι υπέρ. Αποχές δεκτό. 205. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 206. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές δεκτή. 207 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 208 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 19 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 211 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 213. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.15. Ψηφίστε παρακαλώ. Ζητήθηκε λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.15. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. 217. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 221 υπέρ κατά αποχές δεκτή 222 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή ...227 πλέον. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 228 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 228 ψηφίστε παρακαλώ πέρας της ψηφοφορίας δεκτή Τώρα έχουμε τη συμβιβαστική παρήθμη 29, έχουμε τρία τμήματα εδώ κατά διέρεση ψήφο. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό και το τρίτο τμήμα. Περνάμε συνεπώς στην 2.29, Howitt. Ποιοι είναι υπέρ της 229, ποιοι είναι κατά, αποχές δεκτή. 230, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 231, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 232, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ κατά αποχές δεκτή 235-36 από κοινού ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές δεκτές η συμβιβαστική 1 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα της 21 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Περνάμε τώρα στην 2.43 υπέρ, κατά, αποχές. Μόνο τέσσερις ψήφισαν τώρα. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί 2.43 ηλεκτρονικός έλεγχος πλέον. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 2-4-4, 2-44. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2-46. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. 250 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 250. Vediamo la votazione. Approvato. Λοιπόν, δεκτή 250. Συμβιβαστική 22. Συγγνώμη πρόεδρε, όπως και στον προηγούμενο συμβιβασμό, είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας 6. Εμείς συμφωνήσαμε επί της αρχής και περιλαμβάνεται η συμφωνία στην συμβιβαστική 23 μετά από την πρόταση του ΕΛΚ αλλά υπήρξε μια διαφορετική ε, προφορική τροπολογία από πλευράς της συντηρητικής ομάδας ε, και διαφωνούμε με αυτή. Συγχωρείτε, ε, και εμείς συμφωνούμε με αυτή την αντίρρηση. Vuoi oggetto sommernamente Bene, allora ad non lo votiamo Λοιπόν, ε, περισσότερο από όσο χρειάζεται δεν ψηφίζουμε. Λοιπόν, τη θέτουμε σε ψηφοφορία ως έχει τη συμβιβαστική 22, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 254, βερσία Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Επαναλαμβάνω, 254 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η 254. Περνάμε στην 2.57. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Με προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα τις ψηφίσουμε από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 2.60. Τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 264. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. 265. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 269 και 270 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτονται. 2.71. Α, θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 2.69-2.70. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 24. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. Τώρα στην 276. Ποιοι είναι υπέρ της 276. Κατά. Αποχές δεκτή. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 280. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 281 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 25 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.85 τώρα με προφορική τροπολογία υπαρίθμο 8. Scusate, io abbiamo un problema sulla lista di voti. Eccolo qua però non c'è l'emendamento orale. C'è un emendamento orale no? Allora, eh, Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή σύγχυση, στους, υπάρχουν διαφορές στους καταλόγους εδώ. Ψηφίζουμε τώρα την 285 με την προφορική τροπολογία 8. Λοιπόν, από κοινού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Τώρα συμβιβαστική 26. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 287, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 287 Σόλτς. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας δεκτή. 288 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 27 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 286 Α, όχι. 2.93 διορθώνει ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 2.93. 2.94 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2.95 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2.96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.98 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.99 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.99 300 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 301 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 302 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές δεκτή 306 υπέρ ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος για την 304 ψηφίζουμε παρακαλώ την 304 Γιαννάκου ψηφίστε παρακαλώ Πέρα της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή η 307. 306. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 306. Ψηφίστε παρακαλώ. Έχετε αρχίσει και κουράζεστε, αλλά αν δεν βοηθήσετε δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις τέραστη της ψηφοφορίας. Απερίφθη με μία ψήφο μόνο. 307. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 313. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 314 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 315 υπέρ. Με προφορική τροπολογία η 315 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 317 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 320 ποιοι είναι υπέρ αν θέλετε ε, να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, αλλά κάθε φορά αν ψηφίζουν μόνο τέσσερις, πώς να καταλάβω. Λοιπόν, για την 317 ηλεκτρονικός έλεγχος, 317. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 320 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή 322 Α, είναι τεχνικής φύσεως. Περνάμε στην 324. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν, απορρίπτεται. 323. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 323 παρακαλώ. Ψηφίστε. πέρα της ψηφοφορίας. Τρία 25 παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ της 325. Κατά. Αποχές δεκτή. 328 ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 326 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τώρα ψηφίζετε κανονικά, μπράβο σας. 329 με προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Α, κοιτάξτε, πρέπει να ψηφίσουμε και την 327. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ της 327. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν δεκτή. Περνάμε τώρα στην 329 με προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απορρίπτεται. 330. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και πάλι. 3.30, Άρχεται η ψηφοφορία για την 3.30. Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή η 3.30. Τώρα 3.32. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φτάνουμε στο τέλος ε, συνάδελφοι. 3.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.33 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. 3.34 ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτή. 18 ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δε, απορρίπτεται 27 υπέρ Αζητήθηκε ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26. Ψηφίστε παρακαλώ. 26. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή 26. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 33 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Λοιπόν, οι δύο τώρα, ποιοι είναι υπέρ της δύο, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 4 υπέρ Ζητήθηκε κάποιος έλεγχος. Αν θέλετε να ζητήσουμε από την 4 μέχρι τη 17 να ψηφίσουμε ομαδών. Λοιπόν, λοιπόν φαίνεται ότι αυξάνεται και η κούρα και η καλή θέληση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, όλες δεκτές. Πάμε στη συμβιβαστική 30. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Deve 2, deve 8, deve 9. Αν μπλοκ, deve 2, 8, 9 και 14. Αν συμφωνείτε. Μέχρι τα 14. ποιοι συμφωνούν. Ναι. Ε, Κατά αποχές. Τώρα οι 15. 15 υπέρ κατά έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την DEV 15. Vi chiedo di votare. Mancano due colleghi. Tu. Chiusa la votazione. Απορρίπτεται. Allora, fam 1 chi è a favore? Chi è contrario? Φαμ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα στη Συμβαστική 31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 31. δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 31, μη σας παρασύρει εδώ ο συνάδελφος Πάσκου, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. No, era 4 e 5. 4 e 5 insieme. Allora... 4 και 5 μαζί, λοιπόν. Φαμ 4 e 5 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Check for the second part of compromise number 31. Check the four and five? No, second part. Second part. Questo. Ah, la seconda parte del Seconda parte del 31. Allora, torniamo indietro. Πάμε πίσω. Συμβιβαστική 31. Να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα γιατί ζητήθηκε με ηλεκτρονικό έλεγχο. Εγκρίνεται. 4 και πέντε έχουν απορριφθεί. Και πάμε... Φαμ 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 με 14 από κοινού. υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Συνάδελφοι, ψηφίστε γιατί είναι δεν ψηφίσατε. Ε, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Allora, Από κοινού τώρα. 17, 19, 20 και 21. Εάν συμφωνείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 22, eh, sempre me per favore. No, 22. Allora, 22, chi è a favore? 22 υπέρ, κατά. Αποχές, ε, ε, απορρίπτεται. 23, 24, 27, 29 και 32 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 33 και 34 μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι. Χωριστά. 34 υπέρ. Ε, 33 με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Υπέρ. Κατά. ψηφίζουμε λοιπόν. Εντάξει. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία, συνάδελφοι. Ευχαριστώ.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 colleghi, we have to continue. Colleghi, vi prego un attimo di silenzio, dobbiamo continuare i nostri... Παρακαλώ ησυχάστε συνάδελφοι γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Allora, punto 18, definizione di una nuova cooperazione. Σημείο 18 συνεργασία για την ανάπτυξη με την Λατινική Αμερική. Και έχουμε τον Ρικάρντο Κόρτες Λάστρα. Αρμόδιο επί της ουσίας. Τέσσερα λεπτά η εισηγήτρια. Γιατί έχουμε και άλλα να δούμε μετά. Mr. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή ΔΕΒΕ ζήτησε από την Επιτροπή μας μια γνωμοδότηση για την έκθεση ιδίας ε, πρωτοβουλίας ε, για τον ορισμό μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής με τη Λατινική Αμερική. Στόχος είναι να συνεισφέρουμε στην διαδικασία διαπραγματεύσεων του επόμενου μέσου ανάπτυξης και συνεργασίας ε, και το πλαίσιο 2014-2020 και να προτείνουμε νέους διάβλους ε, συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής κύριος στόχος της Επιτροπής μας είναι να δώσει κάποιες κατευθύνσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική ε, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής. Από πολιτική σκοπιά μεγάλη σημασία έχει η θέση ενισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για να βρει τη δική της φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος στόχος της πολιτικής αυτής ορίζεται στο άρθρο 208 της συνθήκης είναι μείωση και μακροπρόθεσμα εξάλληψη της φτώχειας. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η συνοχή παίζει ένα βασικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Είναι πλέον νομική απέτηση και για την υπατιακό πρόσωπο και για την Κομισιόν. Στο σχέδιο τονίζω τη σημασία της ενίσχυσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και την ανάγκη να αναπτυχθούν νέες μορφές συνεργασία με χώρες ανερχόμενε και μεσαίου εισοδήματο μέσω του μέσου αναπτυξιακή συνεργασία και του νέου μέσου εταιρική σχέση. Επιπλέον τονίζω την ανάγκη ενίσχυση της συνεργασία των δύο περιοχών για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ειδικά των δράσεων κατά της φτώχειας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής ένταξης σε περιθωριοποιημένων ομάδων. Είμαι πεπισμένη πως οι αλφασίγμαχοί που στοχεύουν ε, στην παγκόσμια συνεργασία, δηλαδή ο υπαριθμόν 8, θα πρέπει να στοχεύουν στη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Και έτσι θα υπάρχει μια νέα στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ε, χωρών αυτών επίσης ή ο στόχος 86.2 ε, αφορά τρεις στόχους ε, το Μεξικό, την Βραζιλία και την Αργεντινή ενώ ο ΑΣΧ 20 μπορεί να είναι δυνατότητα να βρούμε κοινά κοινό τόπο για να υπάρξει μια συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Στο σχέδιο μου τονίζω επίσης την συνέργεια που μπορεί να υπάρξει από συνολικές συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφόρων υποπεριφερειακών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό ζητάω ένα όραμα συνεργασίας ε, των δύο χωρών αυτών του πλανήτη σε σχέση με την 7η ε, συνέλευση Eurolat που θα πραγματοποιηθεί στη Χιλή τον Ιανουάριο του 2003. Υπογραμμίζω τη σπουδαιότητα τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνω την έμφαση, με έμφαση την έλλειψη μιας ολοκληρωμένη ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στηριξη συνεργασια συνεργασίας Νότου-Νότου και την απουσία σαφών κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συνεργασία Νότου-Νότου και τη διαπεριφερειακή σύνδεση. Τονίζω λοιπόν την ανάγκη επέκταση του πολιτικού διαλόγου με τη Λατινική Αμερική σε διαφορετικά επίπεδα. Τώρα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους που συνεισέφεραν στην προετοιμασία του σχεδίου γνωμοδότησης και κατέθεσαν τροπολογίες. Προσθέτουν σαφή προσθέμενη αξία στο κείμενο και άρα υποστηρίζω τις περισσότερες από αυτές. Υπάρχουν 19 τον αριθμό συν 8 προφορικές τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης και εγώ ίδια έχω καταθέσει 4 τροπολογίες γιατί σύμφωνα με τους κανόνες ε, είναι περιορισμένος ο αριθμός των λέξεων καθώς οι τροπολογίες καλύπτουν διαφορετικά ζητήματα προτείνω να τις ψηφίσουμε μία-μία χωρίς συμβαστικές τροπολογίες και θα ήθελα να επισημάνω κάποιες προβληματικές τροπολογίες με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Πρώτα απ' όλα η υπαριθμόν 11 ε, της κυρίας Λούνατσεκ που προτείνει ε, αν διαπραγμάτευση συμφωνιών με τη Λατινική Αμερική. Δεν συμφωνώ με αυτό καθώς γίνονται ήδη διαπραγματεύσεις και έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια καλή ισορροπία για τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Το ίδιο αφορά και τροπολογία 12 ε, του συναδέλφου Βίλι Μάιερ. Επίσης δεν συμφωνώ με την τροπολογία 5 του Βίλι Μάιερ που υπογραμμίζει πως η καταπολέμηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας πρέπει να παραμείνει βασικός ε, στόχος της ε, στρατηγικής αναπτυξιακής συνεργασίας και με κάνει λόγο για κοινωνικό κράτος και τέλος τροπολογία 10 και με αυτή δεν μπορώ να συμφωνήσω καθώς μιλάει για το ότι καλωσορίζουμε την ε, ύπαρξη περιφερειακών μηχανισμών ολοκληρώσει όπως η ΑΛΜΑ που είναι επίμαχη νομίζω πως και αυτή την τροπολογία δεν μπορώ να την υποστηρίξω τέλος Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να ε, έρθουν την ερχόμενη εβδομάδα για την ψηφοφορία 27 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Ανάπτυξης 24 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μενέντες ε, Ντεβάλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Bueno, en primer lugar quisiera eh, felicitar a la la señora Andriquiene,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 λόγω ε, ενός προβλήματος που υπήρξε σε επίπεδο πληροφορικής οι θέσεις μας δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν αλλά διόρθωσε η γραμματεία το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συνεργατία της με τη Λατινική Αμερική ε, σε καλύτερο επίπεδο συντονισμού ε, με τις φίλες ε, λατινοαμερικανικές χώρες θα πρέπει και αυτές οι χώρες να προχωρήσουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης την οποία έχουν εμπλακεί παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν μέχρι τώρα. Όταν το πετύχουν αυτό τότε η πολιτική μας συνεργασία με τις χώρες αυτές θα είναι περισσότερο ισόρροπη. Λυπάμαι επίσης γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόταση ε, μεταρρύθμισης των ρυθμίσεων τελών και δασμών δεν λαμβάνει υπόψη τον ε, σημαντικό ρόλο που παίζει η Λατινική Αμερική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στερεί από πολλές χώρες ένα σημαντικότατο μέσο επιρροής. Από την άλλη, η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία όπως και το Περού είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια δύνατη έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια σωστότερη εταιρική σχέση και σε μια συμφωνία εταιρικής συνεργασίας. Από ό,τι φαίνεται το 2015 η Κίνα θα ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πρώτο εμπορικό εταίρο της Λατινικής Αμερικής. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να μας πείσει ότι οι προσπάθειές μας θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον να, μας ξεπεράσει η Κίνα. θα πρέπει παράλληλα να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει η υπογραφή συμφωνία Συμφωνίας Συνεργασίας με το Μερκοσούρ. Αυτό είναι απαραίτητο και για τις δύο πλευρές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια για την κατανόησή της, την ανοχή της και τη συγχαίρω για τη δουλειά την οποία επετέλεσε. Ο κύριος Σαλαφράνκα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μια πολύ βαθιά κρίση και άρα η στρατηγική συμμαχία που είχαμε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, είναι και τις ε, οι είναι πάρα πολύ σημαντικές καθώς μιλάμε για το 1 τρίτο των μελών του ΟΗΕ και αυξάνεται έτσι και το παγκόσμιο ΑΕΠ. Ο κ. Ζελβάλε μίλησε για τις σχέσει μας με μονομενες χώρες με τη Λατινική Αμερική, αλλά πρέπει να έχουμε και μια συνολική στρατηγική για τις ε, χώρες αυτές και διάφορες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Προφανώς η πολιτική Λατινικής Αμερικής είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά η πολιτική μου ομάδα ανησυχεί για το ότι κάποιες χώρες μεσαίου μεγέθους στη Λατινική Αμερική δεν συνεργάζονται πλέον με το μέσο ανάπτυξης της ε, περιοχής. Ελπίζω με την ε, την ομοδότηση αυτή η Επιτροπή μας να αναγνωρίσει την ε, σημασία και να πείσει αυτές τις χώρες για τη σημασία της συνεργασίας μαζί μας. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ε, θα ήθελε να προσθέσει κάτι η ίδια. Ωραία, ευχαριστούμε. Σας πενθυμίζω πως η ψηφοφορία είναι στις 27 Μαρτίου. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση για την πρώτη διακοινοβουλευτική συνάντηση με τη Μιαμάρ που έγινε στη Μαλαισία των αρχές Μαρτίου του 12. Σας δίνω αμέσω το λόγο να μας μιλήσετε για τη συνάντηση αυτή που έγινε στη Ραγκούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λέει ο κύριος Γκέμπελς, σαν αντιπρόεδρος, πρώτος αντιπρόεδρος, αντικαθιστώ τον πρόεδρό μας, τον Βέρνα Λάγκεν, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποστείλει μια διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στη χώρα της Μιανμάρ. Και αυτό μετά από το σχετικό άνοιγμα του καθεστώτος, ε, το οποίο ακολουθεί ο νέος πρόεδρος Φανξέγκ. Δεν θα ήθελα να απαριθμίσω όλες τις συνεδριάσεις τις οποίες είχαμε. Συναντηθήκαμε φυσικά με τον πρόεδρο της χώρας, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο των δύο σωμάτων, συναντηθήκαμε με πάρα πολλούς υπουργούς και κυρίως είχαμε την δυνατότητα να συναντήσουμε για πάνω από μία ώρα την κυρία Αουνσουνκή, η οποία όπως γνωρίζετε όχι μόνο έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έχει πάρει επίσης και το βραβείο Σακχάροφ. Δώσαμε λοιπόν στη Λέβη Αν Σουν Κιμ, μεταφέραμε μια πρόσκληση του Μάρτιν Σούλτς έτσι ώστε να έρθει ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να παραλάβει το βραβείο της επίσημα. Θα ήθελα εδώ να πω ότι οι αρχές της Μιαμάρ έχουν εμπλακεί πλέον σε μια διαδικασία η οποία θυμίζει λίγο την σοβιετική περεστρόικα, την περεστρόικα Γκορμπατσόφ, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Πρώτα προχώρησαν στην εκλογή ενός κοινοβουλίου, κοινοβουλίου που αποτελείται από μια μορφή γερουσίας και ένα βουλευτήριο. Οι εκλογές αυτές δεν ήταν βέβαια και πάρα πολύ δημοκρατικές, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, ο στρατός κατέχει το 25% των εδρών και στα δύο κοινοβουλευτικά σώματα. Και ταυτόχρονα το λεγόμενο κυβερνητικό κόμμα κατάφερε να πάρει περίπου το 80% των υπολείπων εδρών. Και αυτό γιατί γιατί το κόμμα της κυρίας Σάουν είχε περάσει σε μποϊκοτ αυτό, σε μποϊκοτάζ αυτών των εκλογών. Ε, δεν πήρε μέρος στις εκλογές αυτές. Από τότε φαίνεται ότι υπήρξε μια κάποια γυτνίαση ανάμεσα στη Λέδη Αουνξούκη και τον πρόεδρο Φαν Σάνγκ. Διότι... Λοιπόν, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το άνοιγμα αυτό. Απελευθέρωσε 6.000 πολιτικούς κρατουμένους η κυβέρνηση και προσπαθεί να προχωρήσει σε υπογραφή συνθήκης ειρήνης με κάποιες μειονότητες της χώρας οι οποίες βρίσκονται σε, ένοπλο, σε ένοπλη σύγκρουση με την κεντρική κυβέρνηση εδώ και 60 χρόνια. Υπήρξαν κάποια πρώτα βήματα, βέβαια δεν έχει τίποτα ολοκληρωθεί. Πάντως, την 1η Απριλίου θα γίνουν νέες εκλογές για την κάλυψη 48 θέσεων. 40 θέσεων για την κάτω βουλή, το πιο σημαντικό σώμα δηλαδή, και 8 ε, εδρών για την άνω βουλή. Αυτές οι 48 θέσεις χειρεύουν μετά από την αποχώρηση των κομμουνιστών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που έγιναν υπουργοί κάποιοι από αυτούς και γι' αυτό χρειάστηκε λοιπόν να γίνει αυτός ο συμπληρωματικός γύρος. Η κυρία Χάν Σουν Κι είναι και η ίδια υποψηφία και το κόμμα της έχει υποψήφιους σε 48 εκλογικές περιφέρειες όπου θα καλυφθούν οι χειρεύουσες έδρες. Εκεί φυσικά και το κυβερνητικό κόμμα αλλά και άλλα κόμματα έχουν κατεβάσει υποψηφίους. Μας έλεγε η κυρία Αγξουνκή ότι οι εκλογές αυτές θα είναι αρκετά ελεύθερες γιατί θα παρατηρηθούν και από τον διεθνή παράγοντα και αυτό το οποίο έχει σημασία να παρατηρήσουμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων που είχαμε είπαμε γιατί δεν θέλατε μέχρι τότε ε, ξένους παρατηρητές. Την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε να υπάρξουν παρατηρητές από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ασιατικές χώρες. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε μια τέτοια αποστολή παρατήρησης χρησιμοποιώντας τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Πάντως θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την πρόσκληση του καθεστώτος της Μιανμάρ. Το πιο εχμηρό πρόβλημα είναι ότι η Μιανμάρ δεν είναι μια τέλεια δημοκρατία, όχι. Αλλά με τις εκλογές και με την διασφαλισμένη ίσως εκλογή της Λέδη Σανσουκή και ενός μεγάλου αριθμού ίσως των οπαδών της θα δημιουργηθεί μια νέα εσωτερική αντιπολίτευση η οποία ελπίζω να λειτουργήσει θετικά. Χωρίς τη σουνκή υπάρχουν 161 ε, πολιτικοί κρατούμενοι πάντα στις φυλακές. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε αυτοί οι 161 πολιτικοί κρατούμενοι να απελευθερωθούν. Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως είναι το θέμα των κυρώσεων που έχει θέσει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ εις βάρος του προηγούμενου καθεστώτος. Από ό,τι νομίζω, και αυτή είναι η γνώμη μου και όλων των πρέσβεων, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήσαμε επτόπ ή στην Ταϊλάνδη, θεωρούν ότι οι κυρώσεις αυτές δεν επηρέασαν τίποτα ουσιαστικά και δεν ενόχλησαν το καθεστώς των στρατηγών. Ο προηγούμενος πρόεδρος οικοδόμησε μια νέα πρωτεύουσα που μοιάζει λίγο με το παλάτι του Τσαουσέσκου στην Ουγγαρία, αλλά στο πιο παρανοϊκό ακόμα. Είναι μια πρωτεύουσα με μέγαρα, παλάτια, υπουργεία και κάποια σκόρπια ξενοδοχεία μέσα στην άγρια φύση που συνδέονται όμως από τεράστιους αυτοκινητοδρόμους, αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στο κοινοβούλιο, που ε, αυτοκινητοδρόμους με 10 λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε πλευρά. Αυτό δείχνει ότι τελικά οι στρατηγοί είχαν πάντα χρήματα και για την οικοδόμηση και για τις αγορές όπλων. Εμείς επιβάλαμε απαγόρευση εμπορίας όπλων με τη χώρα αυτή, αλλά με κάθε διευκόλυνση μπόρεσαν να αγοράσουν όπλα από την Ινδία, από την Κίνα και από πολλές άλλες χώρες. Το εμπάργκο επίσης για την πώληση των πολιτήμων λίθων δεν έδωσε τίποτα. Εκτός Εκτός ίσως από αυτά τα οποία κάναμε για την υφαντουργία της Μιανμάρ, η οποία δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από το σύστημα των γεννητευμένων προτιμήσεων, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ποσοστώσεις, και από 400.000 κόσμο που ασχολιόταν με την υφαντουργία τώρα έχουν μείνει μόνο 80.000. 320.000 Βιρμανές έχουν πλέον χάσει τη θέση εργασία τους λόγω των εκστρατιών που οργανώσαμε εμείς και οι α, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γιατί υποτίθεται ότι έκαναν καταναγκαστική εργασία οι γυναίκες αυτές οι οποίες πάρα πολύ απλά απελήθησαν. και μάλιστα υποστηρίζουν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί ότι η μοναδική άλλη διέξοδος των γυναικών της υφαντουργίας είναι η προσφυγή στην πορνεία. Ε, πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν πρακτική, να επιτρέψουμε στη χώρα να ανοικοδομηθεί και η αναγενόμενη οικονομία της χώρας να μην μείνει μόνο στα χέρια της Ταϊλάνδης, του Χονγκ Κόνγκ, της Νότιας Κορέας και του Βιετνάμ και ίσως της Ινδίας. Είναι παρόντες αυτοί όλοι, ε, η ελάχιστη φαντουργία που παραμένει είναι στα χέρια τους, μόνο μία ευρωπαϊκή επιχείρηση έχει συμφέροντα εκεί και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξουν ε, πιο τακτικές οικονομικές συναλλαγές με τη χώρα αυτή, όχι μόνο σε επίπεδο πετρελαίου, όπου η Total και η Αμερικανική Σευρών πάντα ήταν εκεί και πάντα έδιναν χρήματα στους στρατηγούς και στο καθεστώς τους. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Σας θυμίζω ότι ο Νορβηγός Υπουργός θα έρθει στις 11 και 20. Και γι' αυτό έχει το λόγο η συνάδελφος Λόχ Μπίχλερ. Και μετά η συνάδελφος Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη διάσκεψη των Πρόεδρων που μου έδωσε τη δυνατότητα ως ε, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πάω στην αντιπροσωπή αυτή. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκέμπελς, αλλά με τις τρεις αυτές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, οικονομική, πολιτική και τη σύγκρουση, θέλω να μείνω στην ε, πλευρά της ε, δημοκρατίας. Εντάξει, τα οικονομικά είναι άθλια, ξέρουμε πως 95% ε, του πληθυσμού δεν έχει ρεύμα, υπάρχει υποσυτισμός των παιδιών. Τώρα για τα πολιτικά, ναι, δημιουργήθηκε ένα κοινοβούλιο. Προσπαθούμε να, να δημιουργήσουν δημοκρατικές δομές υπάρχει ένα σύνταγμα του 2008 που δίνει όλα τα δικαιώματα στο στρατό έχει τα δικά του δικαστήρια που υπερέχουν των πολιτικών δικαστηρίων σε καταστάσεις ε, έκτακτης κατάστασης. Όλοι οι υπουργοί πλην ενός του Υπουργού Εμπορίου ήταν ε, πρώην στρατιωτικοί με τον οποίο δεν μπορούσαμε ε, να διαπραγματευτούμε καλά, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση γιατί ξέρετε πως έχει και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ε, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς. Οπότε ξέρετε πως και εντός του στρατού υπάρχουν οι σκληροί και οι μεταρρυθμιστές και τώρα θα δούμε πως θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις γιατί θέλουν βεβαίως να διατηρήσουν τα προνόμια τους και τη δύναμή τους. Οπότε η μάχη αυτή, ε, η διαμάχη μεταρρυθμιστικών και σκληρών είναι κάτι το ενδιαφέρον. Βεβαίως ε, ομολογούν συχνά πως δεν έχουν τη γνώση να προχωρήσουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχετίζονται με την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων αφέθηκαν ελεύθεροι πάρα πολλοί, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Επίσης ε, επιτράπηκαν περισσότερα ελεύθερα ΜΜΕ, αυτό είναι θετικό. Επίσης ε, οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι δεν λαμβάνουν βίζα και αναγκάζονται να πάνε εκεί ως τουρίστες υπάρχει νόμος που επιτρέπει τη δημιουργία συνδικάτων και αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχει καταναγκαστική εργασία, όχι ε, ε, στην υφαντουργία, όπως είπε ο κύριος ε, Μαγίλς, αλλά Γενικώ είναι η μόνη χώρα η οποία έχει καταδικαστεί από τον ILO για αυτό το λόγο η Μιανμάρ. Ειδικά οι μειονότητες εργάζονται καταναγκαστικά υπέρ του στρατού. Υπάρχει και Εθνική Επιτροπή Συμφιλίου που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανεξάρτητη. Αυτό είναι θετικό. Τέλος για τις εθνοτικές συγκρούσεις, ναι, είναι εξωσημείωτο και η νορβηγική κυβέρνηση που θα ακούσουμε σε λίγο τον Υπουργό της στηρίζει την διαδικασία αυτή, αλλά πρέπει να πούμε πως στη σκληρότερη ε, σύγκρουση στην περιοχή κάρεν δεν έχει σημειωθεί πρόοδος και από ό,τι ακούμε από όταν φύγαμε εμείς δεν είναι θετικά τα πράγματα. Οπότε από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι νωρίς για να μιλήσουμε για άρση των κυρώσεων. Πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και να φροντίσουμε ε, και να σημειώσουμε πως ε, κατάβαση του πυρός υπάρχει με μία μόνο εθνοτική ομάδα, όχι με τις υπόλοιπες. Αλλιώς δεν φαίνεται να έχουν επιτύχει κυρώσεις. Ζητώ από την κυρία Γκόμες να είναι πάρα πολύ σύντομη γιατί μας περιμένει ο υπουργό έξω από την πόρτα. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η χώρα εδώ και καιρό. Ναι, ναι. συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία Λοχμπίλερ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία του ανοίγματο χωρίς να έχουμε αμφιβολίες πως μιλάμε για δημοκρατία και τέτοια. Είναι μια αργή διαδικασία, αλλά πρέπει να την ενθαρρύνουμε. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να παρατηρήσουμε τις εκλογές χωρίς ταυτόχρονα να εφαρμόσουμε τις ε, δικές μας προδιαγραφές ε, και δεν μπορούμε να τι εφαρμόσουμε στις εκλογές 1 η Απριλίου γιατί τώρα ήρθε η πρόσκληση και είναι προβληματική όλη η κατάσταση οπότε ίσω μέσω των πρεσβειών ίσως μπορούμε κάτι να κάνουμε αλλά δεν μιλάμε για αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω δεν πρόκειται και για δημοκρατικέ εκλογέ. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε πω τουλάχιστον θα υπάρξει κάποιο άνοιγμα και συμφωνώ πω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην χάσουμε τα μέσα που έχουμε και να σκίσουμε ε, κάποια πολιτική υπό όρους. Άρση τώρα των εμπορικών κυρώσεων. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές. Αλλά να το συνδέσουμε με σαφείς όρους για τις δικές μας εταιρείε. Γιατί μιλάμε για πολύ πλούσια χώρα όσον αφορά το πετρέλαιο και τα ορυκτά. Οι δικές μας εταιρείε λοιπόν πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και κατά την απόψή μου πρέπει να παραμείνουν οι στοχευμένες ε, κυρίως κατά των τύπων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την έλλειψη κινητικότητας ε, στην πολιτική σκηνή και τα ανθρώπινα δικαιώματα να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι ειρηνική συνεννόηση με τις εθνοτικές ε, μειονότητες κτλ. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να φανούμε έξυπνοι. Να μην χάσουμε τα εργαλεία που έχουμε. Μέτρα σύγκρισης και πολιτική υπό όρους. Ε, δύσκολα πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν. Η Ευρώπη κοινωνία των πολιτών εκεί πέρα ξεκινάει και πρέπει να τη στηρίξουμε. Και κάτι άλλο, πρέπει να τους στηρίξουμε με τρόπο ενεργό και νομίζω πως εδώ πέρα ε, ήταν σωστή η Επιτροπή. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών στη Βυρμανία και την κυρία Σάσουση γιατί τη θαυμάζω αλλά το ότι ήταν απομονωμένη τόσα χρόνια περιορίζει κάπως και τις σκέψεις για το τι είναι πιο αποτελεσματικό. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε σε επαφή μαζί της και με τους δικούς της για να προωθήσουμε την διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουμε εδώ τον Νορβηγό Υπουργό εδώ απ' έξω. Έχουμε ήδη καθυστερήσει και μόνο και μόνο για λόγους ευγένειας πρέπει να διακόψουμε και να τον καλέσουμε. Κύριε πολύ ευχαριστώ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 c'è nessuno proprio, eh? No. Sono tutti deputati, non sono di... Bene, colleghi, eh, ci scusiamo con... Eh, Συνάδελφοι, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον ε, Υπουργό για την καθυστέρηση ακόμη μια φορά και να προχωρήσουμε άμεσα στην ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Στόρ, Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας σε σχέση με τον Βορρά, συμπεριλαμβανομένη στη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα τη ενέργεια και των πόρων, των φυσικών πόρων. Η, συνέργαση, η συνομιλία μαζί του είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για την Αραβική Άνοιξη και για όλα τα σημαντικά θέματα. Ε, σε τον καλωσορίζω θερμό και να καλωσορίσω και τον ε, κύριο Πάτο Κομπουγκάλαχερ που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας με τον οποίο επισκεφθήκαμε την Ελβετία μαζί. Ξέρω πως έχετε πολύ γεμάτη μερίσια διάταξη και γι' αυτό σας ευχαριστώ ακόμη πιο πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη του Φεβρουαρίου ο πυργός Στόρ επισκέφθηκε τις χώρες Αραβικής Άνοιξης. Μετά από λίγες μέρες η κυρία Άστον, μαζί με την κυρία Άστον, πήγε στα νησιά Σβάλμπαρ για να συζητήσουν για την, ε, τα θέματα του Βορρά και έπειτα έχουμε και την ομάδα συντονιστών και των δωρητών για τον λαό της Παλαιστίνης. Η Νορβηγία είναι ένα ιδιαίτερα ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας και έχει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο διεθνές προσκήνιο πέρα από την γεωγραφική ή δημογραφική διάσταση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το ρόλο της ε, νορβηγικής κυβέρνησης που προσπαθεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ε, κατάστασης σταθερότητας και ειρήνης στην Μέση Ανατολή και γι' αυτό και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις απόψεις σας ε, για τον Βορρά, για τη Ρωσία, για τα θέματα της ενέργειας και επαναλαμβάνω και για την Αραβική Άνοιξη και ποια πιστεύετε πως θα είναι οι επόμενες φάσεις αυτή της ε, αραβικής επανάστασης στο Μαγκρέπ και όχι μόνο. Πριν να σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο εν συντομία στον συνάδελφο Γκάλαχερ, που και εκείνο θα θέλει να σας χαιρετήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Νορβηγία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι βρίσκομαι στην Επιτροπή σας και συναντάμε και τον κύριο Στόρε, τον Υπουργό Εξωτερικών. Βεβαίω. Χαιρόμαστε για τη στενή οικονομική και πολιτική συνεργασία με την Νορβηγία. Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι εφαρμόζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η νομοθεσία του ΕΟΧ από την Ορβηγία και θέλω να πω πως από όταν ξεκίνησε αυτή η θητεία του Κοινοβουλίου όταν συνάντησα τους συναδέλφους σας και εδώ στις Βρυξελλές και στην Ορβηγία σε τακτική βάση και στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές του ΕΟΧ θα ήθελα λοιπόν να σου πω πως γνωρίζουμε τις, ε, και γνωρίζετε και στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ομολογήσω πως δεν διάβασα την έκθεση ολόκληρη, γραμμή-γραμμή και δεν ξέρω αν την διάβασαν πάρα πολύ, αλλά ε, διάβασα τη σύνοψη. Και θα την συζητήσουμε. Και θα φανεί αυτό και στο ψήφισμα στη μεικτή κοινοβουλευτική ε, διάσκεψη στην Ισλανδία αρχές Μαΐου. Βεβαίω αναφερθήκατε στην Αρκτική και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την Αρκτική. Θα συνεχίσουμε το διάλογο με την Ορβηγία για τα ζητήματα αυτά και σημειώνουμε τη στρατηγική του Νοεμβρίου πέρσι ε, που παρουσιάστηκε Και βεβαίω εμεί ε, έχουμε τη στήριξη της Νορβηγίας για μόνιμο καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Ζήτημα που παραμένει ανοιχτό μετά την ε, περσινή συνεδρίαση στο Νούαρκ ε, στη Ιρλανδία πέρσι και υπάρχει βέβαια και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή πέρυσι τον Απρίλιο στο Όσλο και στο Σβάλμπαρντο που υιοθετήσαμε ψήφισμα για την Αρκτική που καλωσορίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια υφόρο πολιτική για την Αρκτική που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και αναγνωρίζει το ρόλο μας ως ε, υποστηρικτών της έρευνας της Αρκτικής και υποστηρίζει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καθεστώς παρατηρητή. Οι βουλευτές της Αρκτικής θα συναντηθούν ε, και στο Μοντρεάλ και μετά στην Ισλανδία αργότερα φέτος. Τέλος λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος της Νορβηγίας ως ε, τεροκλειδί σε ενεργειακά ζητήματα και βεβαίω επειδή παρέχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά τις ταραχές στην ε, Μέση Ανατολή και την ε, Βόρεια Αφρική είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία στην επίσκεψή σας στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με προσκαλέσετε. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και είναι συμβολικό το ότι ένας υπουργό από την Νορβηγία θα μιλήσει για τη Βόρεια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Και εσείς είστε ανάμεσα στα δύο αυτά βεβαίω. Να πω πως ε, Χαίρομαι που βρίσκομαι στην αίθουσα που έχει το όνομα της καλής μου φίλης Αναλίντ. Κυρίε και κύριοι, αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω είναι ακριβώς να αφαιρθώ στην Αρκτική. Βλέπετε την εικόνα. Η Αρκτική, κατά την ε, άποψή μας, ε, δεν είναι κάτι το γεωγραφικό, είναι κάτι το πολιτικό. Πρόκειται για την διαχείριση του βορρά της ε, Ευρώπης και του πλανήτη. Από την σκοπιά του Βορείου Πόλου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στη σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Καλαχέρη για τις πληροφορίες που δώσατε ε, αλλά θα γνωρίζετε πως τα βασικά στοιχεία αυτής της σχέσης είναι πως ε, είμαστε, έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις η Νορβηγία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολλών συμφωνιών η σημαντικότερη των οποίων είναι η συμφωνία ΕΟΧ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δημιουργεί στους όρους ανταγωνισμού με την εσωτερική αγορά ως πλαίσιο ολοκλήρωσης και συνεργασίας και σημειώσαμε πως η Νορβηγία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και είμαστε πιο σημαντικοί από την Ινδία και την Ιαπωνία. Είναι λοιπόν σημαντική η οικονομική σχέση που έχουμε. Είμαστε κομμάτι της ε, Σέγγεν, των ερευνητικών προγραμμάτων ε, της ΚΕΠΑ και τα λοιπά. Έλεγα επίσης πως η Νορβηγία επομίζεται τις ευθύνες της αλληλεγγύης με τα νέα κράτη-μέλη μέσω των ε, επιχορηγήσεων Νορβηγίας ΕΟΧ που υποστηρίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Χθες υπογράψαμε μνημόνιο με τη Ρουμανία για την περίοδο μέχρι το 2014 και το ίδιο συμβαίνει με τις άλλες χώρες. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2009 έως το 2014 <coughs> για να στηρίξουμε κοινωνικά προγράμματα, κοινωνία των πολιτών, δημοκρατία κτλ. Και θα έλεγα πως καθώς είμαστε μέλος εσωτερικής αγοράς καλωσορίζουμε τους ε, ανθρώπους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Ε, νομίζω κατά κεφαλήν ε, εμείς ε, λαμβάνουμε τους περισσότερους, γύρω στους 300.000 ε, από την ΕΟΧ που ήρθαν πέρσι. Η έκθεση στην οποία αναφερθήκατε είναι 900 σελίδες, ε, οπότε δεν ε, πρέπει να τη διαβάσετε όλοι. Αλλά είναι μια έκθεση που βασίζεται σε έρευνα για τις συμφωνίες μας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίζει το ότι αυτές οι συμφωνίες ήταν αμοιβαία υποφιλής τα 27 χρόνια και είχαμε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Να τονίσω επίσης την ενεργειακή συνεργασία. Συνάντησα το πρωί τον Επίτροπο τον κύριο Έτογκερ. εμεί ε, παρέχουμε 20% του φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωση και θα είμαστε μακροχρόνια αξιόπιστο προμηθευτή και θα συνεισφέρουμε στην ανανεώσιμη πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωση και θα αναπτύξουμε και τι δικέ μα ανανεώσιμε πηγέ. Οπότε, κυρίε και κύριοι, το 2008 είχα μιλήσει σε μια ανάλογη επιτροπή όταν συζητήθηκε η Αρκτική και είναι η βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής μου ταυτόχρονα. Στα 7 χρόνια που κατέχω αυτή τη θέση παρατηρώ πως πολλές κυβερνήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό το θέμα. Πριν από λίγους μήνες μίλησα για αυτό το θέμα στο Χιούστον, στο Τέξας. Έχω μιλήσει στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Όλος ο κόσμος κοιτάει βόρεια γιατί ο Βορράς ενώνει όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαστάσεις σε αυτό. Γιατί λοιπόν είναι αυτή η δική μας η προτεραιότητα. Εμείς ε, αναφέραμε τρεις παράγοντες αλλαγής. Όταν κάθομαι στο γραφείο μου στο Όσλο και κοιτάω αναλυτικά νότια και δυτικά, βλέπω βασικά ένα σταθερό πλαίσιο. Όταν κοιτάω βόρεια, βλέπω πως υπάρχουν αλλαγές. Θα ήθελα να σας αναφέρω. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Το πιο ορατό στοιχείο αυτή φαίνεται στον βορρά. Μόνο 4 εκατομμύρια μένουν στον αρκτικό κύκλο, εντός του αρκτικού κύκλου, αλλά μιλάμε για ε, μια αιστεία γνώσης της κλιματικής αλλαγής. Ανοίγονται νέοι, νέοι ναυτιλιακοί διάβλοι και ε, βεβαίως είναι και ευπαθές το κλίμα. Πριν από δύο εβδομάδες ε, επισκεφθήκαμε με την ε, κυρία Άστον το Σβάλμπαρντ. Δεν υπήρχε πάγος. Το φιόρδο του Σβάλμπαρντ ε, τέτοια εποχή έπρεπε να έχει πάγο, αλλά δεν είχε. Και η μέση θερμοκρασία στο Σβάλμπαρντ ε, ήταν 10 βαθμούς ψηλότερη από ό,τι συνήθως και είχαμε κρύο χειμώνα σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης λόγω των αλλαγών στα ρεύματα και προφανώς η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα, η διάσταση των πόρων και βεβαίως η Ρωσία. Όπως βλέπετε στο χάρτη γειτονεύουμε με τη Ρωσία και η Ρωσία έχει αλλάξει και βρίσκεται ακόμα σε μια διαδικασία αλλαγής. Αλλά να απαντήσω στο θεμελιώδες ερώτημα. Τι νομικό και πολιτικό πλαίσιο έχουμε για να ανταποκριθούμε στο αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτή την περιοχή. Την τελευταία φορά που ήρθα, πριν από τέσσερα χρόνια, Αφιέρωσα λίγο χρόνο στο ερώτημα του εάν υπάρχει νομικό κενό στον Βορρά. Γιατί ως πολιτικοί και κυβερνήσεις πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα νομικά θεμέλια λήψης αποφάσεων. Νομίζω πως πάρα πολλά έχουν αλλάξει από αυτού. Το Μάιο του 2008 τα κράτα οποία βρέχονται από την Αρκτική υιοθέτησαν ε, μια διακήρυξη στη Γρυλανδία όπου δεσμευτήκαμε ε, στο ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για την Αρκτική. Η Αρκτική από νομική σκοπιά δεν διαφέρει από οποιονδήποτε άλλον ωκεανό. Υπάρχει πάγος, αλλά γύρω-γύρω υπάρχουν ε, κράτη που βρέχονται από αυτήν. Ρωσία, Καναδάς, ΗΠΑ, Δανία, Γρυλανδία δηλαδή και Νορβηγία. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ε, με την ανακοίνωση του 2008 της Κομισιόν και με άλλα επίσημα έγγραφα δηλώσεις από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πως υπάρχει ε, ένα νομικό και πολιτικό πλαίσιο στην Αρκτική. Οπότε υπάρχει μια ευρεία συμφωνία επ' αυτού. Γι' αυτό και το τονίζω, δεν υπάρχει κάποιος αγώνας για την Αρκτική. Η, ιδέα είναι, όταν μιλάμε για έναν αγώνα, είναι πως υπάρχει ένα, μια τέρα νουλους και όπου όποιος προλάβει θα αρπάξει ό,τι μπορεί και βεβαίως ε, υπήρχε μια σημαία που κάρφωσαν ε, οι Ρώσοι στο Βόρειο Πόλο. Μα να σα πω πριν από έναν αιώνα το 1911 ένας Νορβηγός έβαλε μια Νορβηγική σημαία στο Νότιο Πόλο. Δεν έγινε Νορβηγικός ο Νότιος Πόλος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα λοιπόν και με τη ρωσική σημαία και δεν παριστάνουν και τίποτα διαφορετικό οι Ρώσοι. Ζητάνε λοιπόν βεβαίως άδειε μεγάλες εταιρείε, αλλά δεν υπάρχει νομικό κενό. Το τελευταίο ζήτημα στο οποίο διαφωνούσαμε με την Ρωσία λύθηκε πέρσι όταν ορίσαμε τα όρια μας στη θάλασσα του Μπάρεντς και υπάρχουν ελάχιστα ζητήματα διαφωνίας περί συνόρων και ορίων στην Αρκτική και αυτό είναι μια καλή αφετηρία κατόπιν Η περιοχή αυτή ε, χρειάζεται γνώση και στην αρκτική μας πολιτική εμείς ε, λέμε πως η γνώση είναι το βασικό μέρος της στρατηγικής μας. Έρευνα, εφαρμοσμένη γνώση για το πώς εφαρμόζουμε τις διαφορετικές ε, δραστηριότητες στο βορρά. Παραδείγματος χάρη στο Σβάλμπαρτ, τα νησιά αυτά, στον 78ο παράλληλο, έχουμε ένα πανεπιστημιακό κέντρο με 350 φοιτητές. Η μισή από αυτούς είναι άλλο δαπή και έχουμε και ερευνητικού σταθμού από χώρε όπω η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία και βεβαίω διάφορα νορβηγικά ιδρύματα. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό από μια σκοπιά ανάπτυξη τη ε, γνώση πάνω στην οποία θα βασιστούν οι αποφάσει. Τι κάνουμε λοιπόν ε, πολιτικά για την Αρκτική. Υπάρχει πέρα από τα κράτη Υπάρχει και το Αρκτικό Συμβούλιο που λαμβάνει σχετικές αποφάσεις. Πριν από 10 χρόνια το μεγαλύτερο πρόβλημά μας ήταν πως κανείς δεν ήξερε τι είναι το Συμβούλιο της Αρκτικής. Σήμερα το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο το ενδιαφέρον. Πέρσι στην Υπουργική Διάσκεψη στην Κρυλανδία συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί μια μόνιμη γραμματεία που θα εδρεύει στην Τρέμψο στην Βόρεια Νορβηγία και θα και εξετάσουμε και αιτήσει για μόνιμους παρατηρητές. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έτσι, μια έτσι την οποία στηρίζουμε. Θα επανέλθουμε ίσως σε αυτό. Να σχολιάσω τώρα για αυτούς τους τρεις παράγοντες αλλαγή, την κλιματική αλλαγή. Λιγότερο από 15% του πάγου ε, στην Αρκτική είναι τώρα νεότερος από δύο έτη, από το 1979 μέχρι το 2006 μειώνεται, ε, έχει μειωθεί κατά 45.000 ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, ο πάγος και όπως σας είπα πρόκειται για ένα εργαστήριο μελέτης κλιματικής αλλαγής και θα προκύψει περισσότερη γνώση και για την IPCC που κάνει παγκόσμιες ε, προβλέψεις. Η γνώση αυτή έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβει πώς αντιδρούν οι ωκεανοί, τα ρεύματα και πώς ε, αλλάζει ο καιρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης συνεισφέρει σε αυτή την έρευνα κατά πολύ ε, να υπάρχουν σημαντικά προγράμματα έρευνα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεύτερο σημαντικό κομμάτι προσβασιμότητα των φυσικών πόρων. Κάποιοι εκτιμούν πως 30% του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί είναι στην Αρκτική. Υπάρχουν επίσης ε, όρεκτα η περιοχή του Μπάρεντς που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η διάβλη ναυτιλιακή. Τώρα μπορεί να πάει κανείς από τη Γιοκοχάμα στο Ρότερνταμ και να γλιτώσει 40% του χρόνου. Όχι όλο το χρόνο, αλλά 6, 8, 10 μήνες ίσως. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση για το τι σημαίνουν αυτοί οι διάβλοι. Τέσσερα πλοία πέρασαν από το βόρειο-ανατολικό ε, πέρασμα το 2008. 38 το 2011. Αλλά 18.000 πλοία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζο, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο. Μόλις ξεκινάμε τώρα και ε, βρισκόμαστε στην αρχή και κάποιοι θα, πούνε, κάποιοι θα περνάνε το καλοκαίρι ε, και θα πηγαίνουν στην Ασία και αντιστρόφως. Αλλά η πιο σημαντική κυκλοφορία θα είναι στην Αρκτική. Είτε μιλάμε για κρουαζιέρες, είτε μιλάμε για ε, εμπορικούς πλώες. Υπάρχει λοιπόν επίσης το υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχει δυναμικό εκεί πέρα για την ανθρωπότητα και ναι, η κλάδοι, όπως η λέξη αυτή, η εκμετάλλευση των ειδών ε, που μπορούν να, να ζουν σε μεγάλα βάθη και μπορούν να περιέχουν πιθανώς φαρμακευτικές ουσίες και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάποιοι υποθέτουν λοιπόν πως όταν υπάρχουν πόροι και διάβλοι θα υπάρχει αγώνας ε, για την εξουσία. Αλλά δεν είναι ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι πόροι δεν αμφισβητούνται και οι γνωστοί πόροι είναι Εντό των ορίων των 200 ναυτικών μιλίων ή της υφαλοκρηπίδα. Εμείς όταν δίνουμε άδειε, ε, είναι ανοιχτέ, ούτω ή άλλω και θα χρησιμοποιηθούν από ε, διεθνεί εταιρείε. Η γενική μου θέση κύριε και κύριοι είναι πως ε, στην Ακτική η Νορβηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μελή έχουν αμοιβαία συμφέροντα. Π.χ. η θάλασσα του Μπάρεντ Ω μια ενεργειακή περιοχή μπορεί να είναι σημαντική για την ε, μακροπρόθεσμη παροχή φυσικού αερίου από την Νορβηγία στην Ευρώπη. Εμεί παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτή την ευθύνη. Η βασική λέξη εδώ πέρα λοιπόν είναι αλληλεξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγία και στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούμε τις εξελίξει για τον ρόλο ε, του φυσικού αερίου στη δική σας τη συζήτηση και για τον ενεργειακό σας χάρτη για το 2050. Ο κλάδος χρειάζεται προβλεψιμότητα και σκοπεύουμε να παίξουμε αυτό τον σταθερό ρόλο. Επίσης έχουμε αμοιβαίο συμφέρον για το μέλλον των πρώτων υλών και την ανάπτυξή τους και παρακολουθούμε τα προγράμματά σας όπως την ε, Ευρωπαϊκή Συνεργασία Καινοτομίας ε, για τις πρώτες ύλες. Οπότε το όραμά μας για την Αρκτική είναι να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες ενώ ταυτόχρονα να διαχειριστούμε τον κείμενο ειρηνικά, υπεύθυνα και με τροπαϊφόρο. Οπότε λέμε χαμηλή ένταση στον, στην Δεν χρειάζεται πουθενά στρατιωτική απάντηση, αλλά θα χρειαστεί μια στρατιωτική παρουσία για να υπάρχει μια τακτική διαχείριση και από πλευράς ναυτιλίας και από πλευράς ε, στρατιωτικής παρουσίας, αλλά χωρί ένταση. Ο τρίτο παράγων, η Ρωσία. 50% τη ακτογραμμή τη Αρκτική είναι η Ρωσία και 50% των πόρων. Πράγματι ε, επηρεάζει την πολιτική της Αρκτικής. Η Αρκτική ήταν ε, θέατρο στο οποίο παίζονταν ο ψυχρός πόλεμος. Ε, εγώ λέω στον κόσμο πως πρέπει πλέον να προσαρμοστούμε στα νέα γεγονότα περισσότεροι έχουν διαμορφώσει μια νοοτροπία ψυχρού πολέμου και δεν πρέπει να ξεχνάμε βεβαίω, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τα νέα γεγονότα. Για την Νορβηγία, που είναι μέλο του ΝΑΤΟ και συνορεύει με τη Ρωσία, βλέπουμε πω στην Αρκτική έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και πρέπει να τα αναπτύξουμε με τρόπο υπεύθυνο. Μία λέξη από αυτού το 1990. Στα σύνορά μας που έχουν μήκο 200 χιλιόμετρα έχουμε ένα φυλάκιο το 1990 λοιπόν είχαμε 5 με 8 χιλιάδες διελεύσεις, ήταν τα πιο κλειστά σύνορα πλήν ίσως της γραμμής ε, Βορείας και Νοτιού Κορέας. Έκτοτε έχουν αυξηθεί. Το 2005 είχαμε 100.000 διελεύσεις, 2011 ε, 200.000 διελεύσεις και τώρα έχουμε πρόβλεψη για 400.000 διελεύσεις. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια φυσιολογική κατάσταση. Το όραμα μας για τις σχέσεις ε, με τη Ρωσία είναι μια φυσιολογική γειτονία αν θα γίνει επί της θητείας μου θα χρειαστεί λίγους χρόνους, αλλά αυτό πρέπει να είναι το όραμα. Απευθεία σχέσεις, ε, επενδύσεις, ε, περιβάλλον, ωκεανή, να διαπραγματευόμαστε στι διαφωνίε ως πολιτισμένα ευρωπαϊκά κράτη. Έχουμε πολλούς ε, Ρώσου φοιτητέ, είναι η μεγαλύτερη ομάδα ξένων φοιτητών στην Νορβηγία και χαράξαμε μετά από 40 χρόνια διαπραγματεύσεων τα θαλάσσια σύνορά μα. Οπότε έχουμε χερσαία σύνορα το 1826 με τη Ρωσία και θαλάσσια σύνορα από το 2011. Οπότε ε, αυτές είναι οι εξελίξεις. Βεβαίω ακόμα ένα πρόβλεπτο το τι θα γίνει στη Ρωσία, τι είδους δημοκρατία θα υπάρξει. Η νορβηγική απάντηση θα είναι συνέπεια, σαφείς θέσεις και μια ανοιχτή προσέγγιση στην εμβάθυνση των σχέσεών μας. Αυτά ως εισαγωγή και βεβαίω θέλω να δεχτώ τις ερωτήσει σα πριν ε, περάσω στο, στο βορρά τη Αφρική μετά. Αλλά θα πω ένα πράγμα. Νομίζω πω όλοι ε, βεβαίω ε, βλέπουμε τα πράγματα από εκεί που βρισκόμαστε. Εγώ μίλησα για αυτό το ζήτημα και στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου πριν από λίγα χρόνια. Και υπήρχε ένα καθηγητή που είπε «Κύριε Υπουργέ, ενδιαφέρον ήταν που μιλήσετε για το βορρά». Για μένα, ξέρετε, βορρά είναι το Σλέσφι Χολστάιν. Και είχε δίκιο. Γιατί ε, αυτό είναι ο βορρά τη Γερμανία. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να σας πω είναι πως αυτό δεν είναι το κέντρο, αλλά είναι ένα νέο κέντρο γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και επαφή σε εμάς ως πολιτικούς και ε, υπεύθυνες δημοκρατίες να το διαχειριστούμε σωστά. Να περάσω τώρα στη Βόρεια Αφρική. Χτες εδώ στις Βρυξέλλες προέδρευσα στην ε, ομάδα Αλχόκ, η οποία ασχολείται με τις ε, δωρήτριες χώρες που ε, προσφέρουν προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι η μοναδική επιτροπή, το μοναδικό φόρουμ, όπου συμμετέχουν ισότιμα το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή. Βοηθούμε την Παλαιστινιακή Αρχή να οικοδομήσει ισχυρές κρατικές δομές, διαρκείς κρατικές δομές και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη να μην σας κουράσω. Υπάρχουν δύο παράλληλες διαδικασίες. Μία εκ των άνω προς τα κάτω που διαπραγματεύεται την λύση τη λεγόμενη των δύο κρατών. Η διαδικασία αυτή ε, εξαρτάται η διαχείρισή της από τα εμπλεκόμενα μέρη και στηρίζεται από το κουαρτέτο και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δυστυχώς η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει, δεν πηγαίνει πουθενά. Οι Ιορδανοί κάνουν προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτή είναι η διαδικασία εκ των άνω προς τα κάτω. Η Νορβηγία ασχολείται με την διαδικασία από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, οικοδομούμε τις δομές που χρειάζονται, διαμορφώνουμε τον σκελετό έτσι ώστε αυτή τη στιγμή υπάρξει κράτος να λειτουργούν ήδη οι θεσμοί και ελπίζουμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι θεσμοί είναι έτοιμοι, τότε θα υπάρξει κράτος και θα είναι έτοιμη η λύση των δύο κρατών. Δεν ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο τώρα. Ανάμεσα στα άσχημα νέα υπάρχουν όμως και πολλά θετικά στον τομέα της οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης και υποδομών. Πέρυσι εδώ στις Βρυξέλλες υπογράψαμε με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών ε, είδαμε ότι οι θεσμοί οι Παλαιστινιακοί έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο ενός σύγχρονου κράτους και μετά από συστάσεις αυτών των τριών θεσμών είπαμε πλέον ότι ε, οι θεσμοί οι Παλαιστινιακοί πλέον είναι σε επίπεδο σύγχρονου κράτους τώρα. Ο τρόπος που αναπτύσσονται δηλαδή οι υποδομές, η παιδεία, οι καθηγητές, η κατάσταση των τραπεζών, νομίζω ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζηλεύουν την σταθερότητα των Παλαιστινιακών πιστοτικών ιδρυμάτων. Είναι ένα υπόδειγμα μελέτης. Ταυτόχρονα οι Παλαιστινιακές αρχές δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη βοήθεια των δωρητριών χωρών. Γνωρίζετε την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Πρωθυπουργό Ελπίζω ότι θα φτάσει κάποια στιγμή η μέρα όπου δεν θα θέλουμε βοήθεια για την Παλαιστίνη. Είναι εργατικοί άνθρωποι, δεν θα έχουν ανάγκη από την βοήθειά μας και τα χρήματά μας θα τα χρησιμοποιούμε αλλού. Όχι ακόμα όμως, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει μια πλήρη οικονομία υποκατοχή. Δεν μπορεί κανείς ε, να έχεις μια οικονομία όπου τα φορολογικά σου έσοντα συλλέγονται από άλλη χώρα και κατά περίπτωση δίδονται στην οικονομία. Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με συνέχεια οδοφράγματα, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και απαγορεύσεις εξαγωγών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πετύχει και η διαδικασία η εκ των άνω. Ανησυχώ λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ποτέ δεν λένε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα στον δημόσιο τομέα. Αλλά είπαν χτες στις Βρυξέλλες ότι αν σταματήσει η χρηματοδότηση αυτών των ιδρυμάτων των Παλαιστινιακών η διαδικασία θα διαραγεί. Και αυτό θα είναι κακό για τους Παλαιστινίους, κακό για τους Ισραηλινούς, κακό για την ασφάλεια της περιοχής. Θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη δωρήτρια χώρα προς την, Ευρωπαϊκή, προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Ακολουθούμε εμείς σαν Νορβηγοί. Ζητούμε λοιπόν Ε, να κάνει πρόοδο και η Παλαιστινιακή πλευρά. Ο Πρωθυπουργό ήδη μα είπε ότι έχει μειώσει την εξάρτησή του από την εξωτερική βοήθεια από 2,5 δις σε 1,5 δις. Έχει προχωρήσει σε διάλογο με τους κοινωνικού εταίρου στην Παλαιστίνη σύμφωνα με αυτά τα οποία γίνονται και στις ευρωπαϊκές χώρες χωρί καμία συνεισφορά από το ΔΝΤ γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο ΔΝΤ. Συνεχίζουμε να λέμε λοιπόν ότι οι Ισραηλινές και Παλαιστινιακές αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν έτσι ώστε οι μηχανισμοί αυτοί να είναι διαφανείς, προβλέψιμοι και λειτουργικοί και διαχωρισμένοι από την πολιτική. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν την οικονομία εκ των έσω. Δεν θα αναφερθώ στα μεγάλα θέματα της Μέσης Ανατολής γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος της Επιτροπής μου αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας, πρέπει να καταδικάσουμε τις ροκέτες, τους, τις δολοφονίες, πρέπει επίσης να είμαστε και κατά των εγκαταστάσεων, των επικισμών των Ισραηλινών, γιατί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές νόμο δίκαιο. Τώρα λοιπόν έχουμε όμως κάποιους κοινού τόσους με τους Ισραηλινούς και πρέπει να τους στηρίξουμε. Τώρα για την Αραβική Άνοιξη, Πρόεδρε, παρακολουθείτε από κοντά όπως και εμείς. Το συμπέρασμά μας είναι ότι για γενιές ολόκληρες θα ζήσουμε τις συνέπειες. Είναι ίσως η πρώτη φορά που υπάρχει μια εξέγευση στην περιοχή αυτή εκ των κάτω από τη βάση. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, τι είδους δημοκρατία τώρα θα αναδυθεί Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο χαρακτηριστικό από τη βάση προς τα πάνω, ενάντια στην κατάχρηση της εξουσίας, ενάντια στον εποτισμό, ενάντια στην διαφθορά και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα έχουμε και περιφερειακές μικρές ιστορίες και σενάρια στο εσωτερικό. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη βία α, καταπιέζοντας τα καθεστώτα τους στην Ιεμένη, στη Λιβύη και και το ίδιο θα συμβεί και στη Συρία φαίνεται ότι θα χάσουν την εξουσία. Οι χώρες αυτές πέρασαν σε μεταρρυθμιστικές, οι χώρες μάλλον που πέρασαν σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες νωρίτερα, όπως το Μαρόκο και εν μέρη την Ισία θα πετύχουν. Ο κοινό παρανομαστή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν φιλελεύθερε δημοκρατίε είναι πώ θα αντιμετωπίσουμε εμεί τι πολιτικέ επιλογέ στο μέλλον για τι χώρε αυτέ. Νομίζω ότι αυτό μας παρουσιάζει πάρα πολλές προκλήσεις. Θυμίζω ότι δεν ξεκίνησε στην Τινησία η Αραβική Άνοιξη, ξεκίνησε στην Αλγερία στα τέλη του 80. Η κατάληξη ήταν καταστροφική. Είχαν ε, εμφύλιο πόλεμο και πάνω από 50.000 νεκρούς. Πώς λοιπόν θα μπορέσει η νέα πολιτική τάξη να αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτό που μπορώ να πω χωρίς να είμαι σίγουρος είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους εμπλέξουμε στις δικές μας διαδικασίες. Εγώ είχα επαφές με κάποια από τα κινήματα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θα συναντηθούμε με αντιπροσωπείες αιγυπτιακές έρχονται σε εμά για να μελετήσουν το δικό μας πρότυπο ε, κοινωνικής πρόνοιας. Ε, δεν μπορεί να αντιγραφεί ένα τέτοιο πρότυπο, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να μοιραστεί τις πετυχημένες εμπειρίες και αυτό μπορεί να το κάνει επιμένοντας και στον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι διαπραγματεύσιμα και εφαρμόζονται σε όλα. Ελευθερία έκφρασης, ελευθερία θρησκευτική, ελευθερία του συνέρχεστε, ισότητα ανδρών γυναικών. Και η διαφορά τώρα από το 1989 στην Αλγερία είναι ότι σήμερα η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί και αν δεν μπορέσουν να διορθώσουν τα οικονομικά προβλήματα είτε θα γίνουν σαν τη Βόρεια Κορέα είτε θα ολοκληρωθούν μεταξύ τους και αν ολοκληρωθούν μεταξύ τους θα πρέπει να διαχειριστούν την οικονομία τους με διαφανή τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και να αναπτυχθούν. Έτσι, έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Τώρα, για την Μιανμάρ, ε, την οποία συζητούσατε πριν πω, την επισκέφθηκα και αυτήν και εκεί πέρα βοηθάμε και ε, είχα και εκεί πέρα την ίδια εντύπωση πως οι στρατηγοί στη Μιανμάρ έχουν μια επιλογή. Είτε συνεχίζουμε και πρέπει να κλείσουμε την πόρτα και να γίνουμε Βόρεια Κορέα ή αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να ανοίξουμε στον έξω κόσμο και να εξυγχρονιστούμε. Αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ο ταξιτζής στο Κάιρο που πηγαίνει τουρίστες στην πυραμίδα, έχει ακόμα, στις πυραμίδες, έχει ακόμα κενέ κούρσε. Αν δεν γεμίσουν τα ταξί και πάμε στι παραλίε, και για να πάμε στι παραλίες θα θέλουμε να αφορέσουμε μπικίνι, ό,τι θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, μόνο τότε θα αναπτυχθεί η οικονομία τη Αιγύπτου. Και δεν θα υπάρξουν επενδύσει σε αυτές τις χώρες αν δεν είμαστε σίγουροι πώ τα λεφτά θα εξοδευτούν σωστά και όχι σε διαφθορά. Ξέρω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ρόλο κλειδί και σας ενθαρρύνω να εμπλακείτε και εμείς θα σας στηρίξουμε. Για τη Συρία νομίζω έχουμε παρόμοια προσέγγιση για τα φρικαλαία γεγονότα. Η Νορβηγία συμμετείχε στην ε, στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Θεωρούν πως δεν είναι κατάλληλη αυτή η λύση για τη Συρία. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του αραβικού συνδέσμου και ενθαρρύνουμε και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οπότε κύριε Πρόεδρε, ε, εδώ θα ήθελα να ολοκληρώσω την επισκόπηση της Βόρειο Αφρικής από τη Βόρεια Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Τώρα θα ακούσουμε τους ε, συνάδελφους. Πρώτος στον κατάλογο η κυρία Γκόμεζ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μια πνοή φρέσκου αέρα από το βορρά και ελπίζω να παίρνετε μαζί σας την κυρία Άστον συχνότερα, όχι μόνο στο βορρά, αλλά και στο νότο, στην Ανατολή. αποφεληθούμε οπωσδήποτε από την ε, προσέγγισή σας και τη διάθεσή σας να αλλάξετε τα πράγματα. Και να πω επίσης ε, πως ε, θαυμάζω την πολιτική αρχών που ακολουθεί η χώρα σας και αυτό το έζησα ειδικά σε μια χώρα αγαπητή σε μένα, στο Τιμόρ, το Ανατολικό Τιμόρ. Ε, παίζει μεγάλη σημασία ακόμα η Νορβηγία στις προσπάθειες που γίνονται για τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Και να σας ευχαριστήσω επίσης για τη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης. Θα έλεγα μόνο πως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν οι ανησυχίες σας, όπως αναφέρατε, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, παραδείγματο χάρη στον αραβικό κόσμο, να τις ε, θέτατε και στους Ευρωπαίους ομόλογους σας γιατί μεγάλο κομμάτι της τωρινής ε, κρίσης ακριβώς σχετίζεται με την απορρίθμιση αυτή που προώθησε τη διαφορά και πολλά από τα προβλήματα που έχουμε τώρα για να ξεπεράσουμε την κρίση και το ότι αισθάνεται ο λαός μας και στη χώρα μου, την Πορτογαλία, σχετίζεται με την αδικία της διαφθοράς και των ανισορροπιών. Και συγκεκριμένα το ζήτημα το να καταπολεμήσουμε τις ε, offshore, τους φορολογικούς παραδείσους. Ελπίζω η Νορβηγία να ηγηθεί και σε αυτό τον τομέα. Τώρα, το ερώτημά μου. Πρώτα απ' όλα. Αυτά τα οποία μας είπατε για την Αρκτική είναι πράγματι ε, πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε πράγματα περισσότερα για τις προοπτικές και τις δυσκολίες που υπάρχουν και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γιατί λέτε μία από τις προκλήσεις είναι η κλιματική αλλαγή αλλά στη ΣΥΠΑ τώρα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας η προεκλογική εκστρατεία είναι κακή λέξη η κλιματική αλλαγή ακόμα και στο προοδευτικό στρατόπεδο ε, δεν ασχολείται κανείς βρίσκονται σε άρνηση. Και η ΙΠΑ είναι επίσης κρίσιμος ε, παράγων στην Αρκτική. Πώς θα βλέπετε λοιπόν τα πράγματα. Μετά η Ρωσία. Ε, τονίσατε τη σημασία της Ρωσίας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να επεκταθείτε λίγο στο πώς βλέπετε την πρόοδο στη Ρωσία. Βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους, διαδηλώνει. Ε, από την άλλη, ο κύριος Πούτιν ε, επανεξελέγει. Πώς βλέπετε τη διαδικασία πολιτικής αλλαγής στη Ρωσία ε, για να ξεφορτωθεί την ολιγαρχία η Ρωσία και πώς μπορούμε όλοι να παίξουμε ρόλο σε αυτή τη διαδικασία και να μην είμαστε αντιπαραγωγικοί. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφέρατε τη Γερμανία και εκτιμώ αυτό το οποίο είπατε χτες συζητήσαμε για το Ιράκ. Και ξέρω πως η Νορβηγία επίσης παίζει ένα ρόλο. για το ζήτημα εκείνων που βρίσκονται στο στρατόπεδο του Ασράφ. Βέβαια, δεν είναι το σημαντικότερο ζήτημα σχέση μας με το Ιράκ, αλλά ε, καμιά φορά επισκιάζει τα άλλα ζητήματα. Το τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να στηρίξουμε το Ιράκ. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι το να δεχτούν οι ευρωπαϊκές χώρες ε, αυτούς τους ανθρώπους που κρατούνται εκεί. Μπορείτε να μας πείτε αν η κυβέρνησή σας μπορεί να συνεισφέρει και σε αυτό. Και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτά τα οποία είπατε για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί εδώ πέρα ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει από την οτροπία αυτή και χαίρομαι με αυτά που άκουσα από εσά. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Πρέπει να είστε λίγο πιο σύντομοι για να αφήσουμε και ώρα για τις απαντήσεις του Υπουργού. Ε, διαφορετικά, άμα τα λέμε απλώς μεταξύ μας, Δεν ωφελεί πολλά. Λοιπόν, ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ε, καλωσορίζω κύριε Υπουργέ στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών μας. Μόλις έμαθα ότι μάλλον επέθανε ο τρομοκράτης της, της Τουλούζης. Ε, απλώς σας το λέω γιατί είδα τώρα εδώ online. Ε, ήθελα να σας ενημερώσω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε όταν υπογραμμίσατε πόσο μεγάλος είναι ο βαθμός ε, ολοκλήρωσης της Νορβηγίας με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Σέγγεν και τη συμμετοχή σας σε προγράμματα. δεν αφορά μόνο εσάς, ή τα περισσότερα κόμματα ή από το κοινό της Νορβηγίας ε, θα είστε τόσο ελκυστικοί ε, τόσο πολύ μάλλον έλκεστε προς τα δω που συμμετέχετε χωρίς ε, να μπορείτε να πείτε να, να πούν τίποτα ε, χωρίς να κινούν ψηφίσματα κτλ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την καλή σας συνεργασία για, με τις πολιτικές της Ένωσης. Όσον αφορά ως εισηγητής μάλλον του Κοινοβουλίου για τον Βορρά αφού άκουσα τα όσα είπατε Βρίσκω ότι συμφωνούν ε, με την έκθεση που συνέταξα ε, μαζί με τους συναδέλφους ε, πέρυσι και είμαι ευτυχής που βλέπω ότι συμφωνούμε. Αν και εκφράστηκαν κάποιες διαφορετικές ιδέες παλιότερα. Αφού δεν είμαστε Ε, μάλλον ε, ε, έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα, σε αναφέρατε διάφορες πτυχές και για μένα είναι πολύ σημαντικός προς αυτό να έχουμε τέτοια στενή σχέση και να έχετε κι εσείς με τη Ρωσία, δεδομένου ότι έχουν το 50% της ακτής της, της ακτογραμμής Ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει συνεργασία σε όλη αυτή την ακτή με τη Ρωσία. Υπάρχουν ίσως τομείς όπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει και όσον αφορά το περιβάλλον και ίσως εδώ θα μπορούσατε κάπως περισσότερο να επεκταθείτε. Είναι σημαντικό όταν υπάρχει συνεργασία με τη Ρωσία να ισχύουν τα δικά σας υψηλά περιβαλλοντικά στάνταρ σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να σας ζητήσω την εκτίμησή σας σε σχέση με την ε, Μέση Ανατολή. Όπως είπατε υπάρχει αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και λειτουργείται ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μήπως θα ήταν λοιπόν σημαντικό αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω να προσπαθήσει να επιτύχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και ενώ συγκεκριμένα άτομα που θα συμμετέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ε, τους υπολείπους να γνωριστούν μεταξύ τους. Έχουμε πολλά, εμείς εισάγουμε, εδώ, φέρνουμε εδώ Παλαιστινίους, Ισραηλινούς, Ευρωπαίους νέους και συναντώνται εδώ. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, αλλά ίσως ε, επιτόπου θα έπρεπε να γίνεται προσπάθεια με τη δική σας συμμετοχή, να ενθαρρύνουμε δηλαδή την ε, Παλαιστινιακή και την Ισραηλινή κυβέρνηση να δεχτούν τακτικές ανταλλαγές νέων μαθητών, ώστε να φύγει ο φόβος και να εξαλειφθεί η αρνητική προπαγάνδα, ή να μην κερδίζει έδαφος στις καρδιές των νέων. Υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε λοιπόν αυτές τις ανταλλαγές και τελευταίο σημείο σε σχέση με την πολιτική ε, παρατήρηση, παράδειγμα που κάνατε το πολιτικό Ισλάμ ξεκίνησε το 79 στο Τεχεράνι, αν και δεν είναι αραβικό, είναι περσικό ε, το Ισλάμ αυτό. Είπατε ε, γιατί η ριζική, η ριζοσπαστική πτέρυγα του πολιτικού Ισλάμ κινείται βασικά από την Τεχεράνη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια τεράστια πρόσκληση αυτή τη στιγμή, ώστε να σταθεροποιήσουμε τις χώρες με βάση τις συγκεκριμένες τους ε, συνθήκες. Εγώ ήμουν από την Τινησία, όπου είμαι σχετικά αισιόδοξο και ήμουν ο κεντρικός παρατηρητής για τις εκλογές εκεί. Αλλά αν δούμε μια τεράστια χώρα όπως η Αίγυπτη, Αίγυπτος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το ερώτημά μου είναι, η διεθνής κοινότητα έχει τη δυνατότητα να πείσει τους ηθήνοντες που είναι σε μεγάλο βαθμό αισθητικοί ώστε να αφήσουν την κοινωνία να αναπτύξει το πολιτιακό της σκέλος και το δημοκρατικό μονοπάτι που θέλει να ακολουθήσει. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Γιάκο Ανσάρη. Ευχαριστώ. Μια χαρά το είπατε. European and Εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις έρευνες που κάνει η Νορβηγία στις αρκτικές περιοχές. Πολύ σημαντική δουλειά και πολύ καλά τα νέα που μας είπατε ότι το Αρκτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει τις δυνατότητές του για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις εγκαθιδρύοντας μια μόνιμη γραμματεία στην Νορβηγία. Γιατί είχαμε προτείνει και εμείς ε, ένα κέντρο ενημέρωσης στη Λαπωνία. Ε, να αναφέρω ότι εμείς ε, Είμαστε και εμείς μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου, αλλά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χάρη στην νέα τεχνολογία έμαθα για μια πολύ σημαντική διάσκεψη ε, που γίνεται σήμερα στην Νορβηγία. Ο αναπληρωτής υπουργό Εξωτερικών ε, μιλάει σήμερα για τη Λευκορωσία στην Νορβηγία. Ε, εντάξει, δεν είναι το θέμα στη Λευκορωσία, αλλά θα ήθελα να σα ρωτήσω για την άποψή σα για τι σχέσει με τη Λευκορωσία. Εντάξει, δεν αφορά, δεν είναι Ρωσία, είναι Λευκορωσία. Οπότε τι άποψη για την τρέχουσα κατάσταση και για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Γιατί για εμάς είναι όλο και πιο δύσκολο να, δούμε κάποιο φως στο τέλος του τούνελ. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες, έφυγε. Αλλά σημειώνω αυτά τα οποία είπε περισσότερο παρατηρήσεις. Ε, έκανε και μια ερώτηση για το στρατόπεδο Άσραφ. Ε, θεωρώ πως θα πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή σύμφωνα με, τη... με αυτά τα οποία λέει ο ΙΕ και τη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρω πως πολλοί που εδώ πέρα, αυτή είναι η απάντησή μου. Λοιπόν, για τον κύριο Γκάλερ. Τώρα, ξέρετε, υπάρχει περιθώριο για όλους για να συνεργαστούν με τη Ρωσία. Αυτό το οποίο κάνουμε μέσω του ΠΟΕ, διάφορους τρόπους ολοκλήρωσης, είναι όλα σημαντικά. Να επισημάνω πως στο Βορρά θεωρώ πως ε, υπάρχει μια περιφερειακή περιοχή, το Συμβούλιο της Θάλασσας Μπάρεντς, το Συμβούλιο της Βαλτικής, η Βόρεια Διάσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Αρκτικό Συμβούλιο, ε, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αλληλεπικαλύπτονται και είναι πολύ ρεαλιστικοί. Αφορούν διασυνοριακά ζητήματα και λύνουν αρκετά από αυτά και η εμπειρία μου σε συνεργασία με τη Ρωσία στο πλαίσιο αυτό είναι καλή. Ασχολούμαστε με, ασχολούμαστε με τους ε, αυτόχθονες ε, πολιτισμό, εμπόριο κτλ, επιστημονική συνεργασία και είναι είναι καλό ε, τρόπο συνεργασία και προσωπικέ επαφέ. Ακούσατε για την άποψή μου για τι διελεύσεις των συνόρων. Κάποιοι ασκούν, ασκούσαν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση πω τα 10 πρώτα χρόνια μετά την πτώση του τύπου του Βερολίνου ήταν μόνο πολιτισμό ε, και ε, προσωπικέ επαφέ και όχι επενδύσει. Αλλά αυτή ήταν η ανάλυση μα τότε. Όταν άνοιξαν τα σύνορα έπρεπε να καλύψουμε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ήταν σαν να έκλεινε μια παρένθεση και έπρεπε να επανέλθουμε στη 18ο αιώνα να δούμε πώς ήταν η σχέση τότε. Εμείς είχαμε στείλει πρώτη πρεσβεία στο Αρχαγγέλσκ τον 18ο αιώνα. Επί... Εμείς δηλαδή ήμασταν υπό κυριαρχία της Δανίας. Κλείσαμε το γενικό προξενείο που είχαμε, που το είχαμε και όταν γίναμε ανεξάρτητοι και αναγκαστήκαμε να το κλείσουμε το 1936 ε, λόγω Στάλιν που έβλεπε παντού φαντάσματα. Πριν από δύο χρόνια ε, γενίασα ξανά προξενείο στο Αρχαγγέλσκ. Επανερχόμαστε λοιπόν σε κάτι το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Για τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές στη θάλασσα του Μπάρεντς είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τη Ρωσία για την υγιεινή και ασφάλεια στις βιομηχανικές δραστηριότητες στη θάλασσα του Μπάρεντς. Είναι δύο ζώνε, αλλά ένα οικοσύστημα η θάλασσα του Μπάρεντ ε, και πρέπει να το δούμε συνεπώ. Για το πολιτικό Ισλάμ συμφωνώ. Αυτό το οποίο είπα εγώ ήταν πω η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε τότε. Άξι μπορείτε να πείτε πώ ε, όλα είχαν ξεκινήσει από την Περσία αλλά το παράδειγμα του Ιράν ε, προκαλεί σκέψη. Εγώ θεωρώ πως μιλώντας με τις νέες αυτές οι δεν πάνε προς τα εκεί. Σκέφτονται Τουρκία και η Ινδονησία ως παράδειγμα αλλά εάν λέει αν δει κανεί βεβαίω και το τι έλεγαν το 79 και 80 Ιρανοί, ούτε αυτοί είχαν προβλέψει την κατάσταση που ακολούθησε. Ναι. Ε, τότε πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτού του ανθρώπου και να απαιτήσουμε λογοδοσία. Ε, δεν είναι μέλλον το να λέμε δεν μα αρέσουν αυτά τα οποία βλέπουμε και σα κλείνουμε την πόρτα. Δεν γίνεται αυτό. Για το συνάδελφο τώρα από τη Φιλανδία. Την συνάδελφο. Χαιρετίζω τη Φιλανδία που εκπροσωπεί τον αρκτικό κύκλο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Πρωθυπουργός Ολίπονεν έθεσε την βόρεια διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάμαι. Τώρα, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρκτικής. Πρώτα απ' όλα, τρία κράτη-μέλη είναι ε, μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία και βεβαίως και εμεί συνδεόμαστε στενά. Και η Ισλανδία, αν μπει, θα είναι τέταρτη χώρα. Αλλά δεύτερον, όταν ήρθε η Λέδη Άστον στο Σφαλμπάρτ, είδαμε εκεί πέρα πως γίνεται σημαντική έρευνα. Και εάν τα ζητήματα της Αρκτική που είναι παγκόσμια, κατά την άποψή μου, ε, τονιστούν περισσότερο στο 8ο πρόγραμμα έρευνα, αυτή είναι μια συνεισφορά της Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εκφράζεται τώρα, στηρίζει τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου της ε, Σύμβασης του ΟΗΕ, όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ενισχύσει ένα σταθερό ε, νομικό πλαίσιο, πολλές από τις, νομικές, ε, πολλές από τις ναυτιλιακές μεταφορές από και προς την Ευρώπη έρχονται. Εγώ ανέφερα το δρομολόγιο Ρότερνταμ και κοχαμα ευρωπη Ευρώπη-Ασία. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε. Ε, για τον κύριο Λίζεκ και τη Λευκορωσία συμφωνούμε με τις ανησυχίες σας ε, και βεβαίω ε, η Νορβηγία ευθυγραμμίζεται με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά μέτρα. Ξέρετε, η Νορβηγία είναι υπέρ της αυστηρής τιμωρίας όσων εγκληματούν, αλλά κατά της θανατικής ποινής. Και είναι κρίμα το ότι υπάρχει θανατική ποινή στην Ευρώπη. Και υπήρξε μια εκτέλεση της προάλλες στη Λευκορωσία. Είναι μια δικτατορία που πρέπει να λογοδοτήσει. Αλλά να αναφέρω ένα συγκεκριμένο τομέα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο Βιλνίος. Που είναι ένα πανεπιστήμιο, μπορεί να το έχετε επισκεφτεί, με φοιτητέ από τη Λευκορωσία που πάνε στη Λιθουανία, στο Βίλνιους, για να λάβουν μια σύγχρονη ε, ποιοτική εκπαίδευση. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι αυτή τη στιγμή πρόβλημα η οικονομική επιβίωση αυτού του πανεπιστημίου. Πρέπει να το βοηθήσουμε. Είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά είναι μια ανάσα για τους νέους να λάβουν ποιοτική εκπαίδευση και να πάνε πίσω στο Μίνσκ και να είναι έτοιμοι για το μέλλον. Οι χώρες ε, του Σκανδιναβικού Συμβουλίου στηρίζουν αυτό το Πανεπιστήμιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν τη σημασία του. Γιατί αν αποτύχει αυτό το πανεπιστήμιο θα είναι ε, ακριβώ το λανθασμένο μήνυμα, αυτό που δεν πρέπει να στείλουμε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την εξαιρετική παρουσίασή του. Καλή επιτυχία εύχομαι στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Very welcome.